από αυτή την επιθυμία, αλλά εν πάση περιπτώσει χαίρομαι που βρίσκομαι στην Προεδρία σήμερα και που έχω εδώ και την Αντιπρόεδρο Κόριν Λεπάς μαζί μας. Στο τελευταίο τμήμα, σήμερα το πρωί, τελευταίο τμήμα της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος για αυτή τη βδομάδα, θα εξετάσουμε το θέμα της νόσου του Αλσχάιμερ και άλλων ε, ασθενειών που προέρχονται από την άνοια. Έχουμε μια έκθεση στην ε, Επιτροπή μας για αυτό το θέμα με την Μαρίζα Μάτιας, η συγγήτρια. Θα ψηφιστεί στην Επιτροπή μας. Τι συζητάμε, σίγουρα η κυρία Ματίας θα μιλήσει για το τι θα γίνει στη συνέχεια. Τα συμπεράσματα της σημερινής συνεδρίασης θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη συνέχεια και πάρα πολύ σημαντικά για να εκπονήσουμε τροπολογίες, να συντάξουμε τροπολογίες και να συμπληρώσουμε και την έκθεση της κυρίας Μάτιας αλλά και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευθύ αμέσω θα αναφερθώ στι σημερινέ μα εργασίε. Έχουμε διάφορα τμήματα. Έχουμε λοιπόν ένα εργαστήριο πρώτα απ' όλα, με πρώτο τμήμα την πολιτική και του θεσμικού εκπροσώπου. Εδώ θα μιλήσει και η συγγήτρια, αλλά και κάποιοι άλλοι. Πρέπει να σας πω ευθύ αμέσω ότι στην ημερήσια διάταξη λέει ότι θα ακούσουμε την κυρία Τσίλα Τσέλτον. Και όλοι περιμέναμε να τη δούμε, να την ακούσουμε. Το 2008 βραβεύτηκε ως καλύτερη ηθοποιός για το ρόλο της στην ταινία Pandora's Box, το κουτί της Πανδώρα, όπου είχε το ρόλο ε, της Νάρσετ και βραβεύτηκε στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Όμως χτες το βράδυ χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο γιατί είχε κάποια προβλήματα. Η κυρία Αρή όμως, που είναι πρόεδρος της Λίγας για το Αλσχάιμερ, της Ένωσης για το Αλσχάιμερ, ήρθε και θα μας πει αυτά που θα μας έλεγε εκείνη, θα την εκπροσωπήσει όσο γίνεται τέλος πάντων και θα μας πει αυτά που θα μας έλεγε η κυρία Τσίλα Τσέλτον. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Και βέβαια η κυρία Τσέλτον παρακαλώ ε, να, στην κυρία Τσέλτον να της μεταφέρετε τις ευχές μας για περαστικά. Εγώ ήθελα πολύ να τη συναντήσω προσωπικά. Πριν από δύο χρόνια δεν θα ξεχάσω το βραβείο που πήρε για τον καλύτερο γυναικείο ρόλο. Παρακαλώ να την ενημερώσετε γι' αυτό και να της πείτε ότι της ευχόμαστε περαστικά. Και γρήγορη ανάρρωση. Κυρίε και κύριοι, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Και με ιδιαίτερη χαρά δίνω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την Μαρίσα Μάτιας, για να μας παρουσιάσει τις δικές της ιδέες και να μας ενημερώσει για την έκθεσή της. Μαρίς, έχεις το λόγο. Thank you, Dagmar. Thank you all for being here. Uh, I'll move quickly to the Portuguese. Okay, okay. Συγγνώμη, αλλά θα μιλήσω πορτογαλικά, αν δεν σας πειράζει. Okay, muito bem. Obrigada a todos e a todas. Ευχαριστώ ε, όλους τους παρισταμένους. Φαντάζεστε τη χαρά που νιώθω που διοργανώσαμε το σεμινάριο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πιστεύω ότι ε, τα θέματα που συνδέονται με την νόσο του Αλτσχάιμερ και συγγενείς ε, νόσους, καθώς ε, και όλες τις σχετικές ανακοινώσεις θα πρέπει να οδηγήσουν σε συσπήρωση όλων, θα πρέπει να μας ανησυχούν όλους. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ με πάγιο τρόπο. Το σημερινό εργαστήριο απηχεί την κοινή εργασία που επιδιώκουμε να κάνουμε στον τομέα αυτό είναι η υποχρέωσή μας να δώσουμε απαντήσεις, να ψάξουμε τις απαντήσεις, γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Θα αρχίσω από το τέλος, να. γιατί μες φορές αυτό χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου. Θα αρχίσω ευχαριστώντας με τις ευχαριστίες προς όλους τους προσκεκλημένους ε, που δέχτηκαν να συμμετάσχουν στο σημερινό εργαστήριο. Να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, που έδωσαν θεμελιώδη υποστήριξη για να υλοποιηθεί το σημερινό εργαστήριο, ε, κυρίως τους συναδέλφους μου που κάθονται εδώ στο Προεδρείο και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μου και την κυρία Ντάκμα Ρογκμέρεντ προφανώς που θα ε, διοργανώσει τη σημερινή συζήτηση. Θα συζητήσουμε σήμερα την έκθεση μου, αλλά επειδή ε, θα παρεμβληθεί και το σεμινάριο, δεν θέλω να χαραμίσω το χρόνο σχολιάζοντας ε, το περιεχόμενο της έκθεσης, το γνωρίζετε εξάλλου. Ε, το σημαντικό είναι να ακούσουμε τις φωνές αυτών που δεν ακούμε συνήθως. Και γι' αυτό προσκαλέσαμε τους επαΐοντες, ε, τα μέλη των οργανώσεων των ασθενών, τους εκπροσώπους ε, των πολιτικών θεσμικών οργάνων, ούτω ώστε να συνταχθούμε όλοι και να επιτελέσουμε μια πλήρη εργασία, την ε, βέλτιστη δυνατή εργασία, ούτω ώστε να δώσουμε την καλύτερη δυνατή απάντηση, γιατί υπάρχουν οι προσδοκίε ε, των πολιτών ε, που ζουν καθημερινά με αυτό το πρόβλημα. Δεν θα μακρηγορήσω, θα ήθελα να σας ακούσω κυρίως, να μάθω από σας και μετά από αυτό το εργαστήρι ε, και στο μέτρο που θα έχουμε ακόμη χρόνο για να συζητήσουμε τη βελτίωση της ε, υποσυζήτησης έκθεσης, ε, θα ακούσουμε και τις δικές σας συστάσεις για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο των εργασιών μας. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε, για να μάθουμε από σας, να συζητήσουμε. αυτά και μένω προς το παρόν. Thank you very Uh, Ευχαριστούμε Μαρίσα. Κατάλαβα αυτά που είπες στα πορτογαλικά. Παρ' όλα αυτά εγώ συνεχίζω με τα αγγλικά. Ξέρω ότι δεν ενθουσιάζονται διερμηνείς από αυτό, αλλά λέω εκ των προτέρων συγγνώμη, λέω μιλήτρια. Αλλά αισθάνομαι ότι έτσι υπάρχει μεγαλύτερη αμεσότητα μεταξύ μας. Ευχαριστώ λοιπόν Μαρίσα. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσουμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ακούσουμε την ε, παρουσίαση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Alzheimer και άλλες ε, ασθένειες και να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για να στηρίξουμε τις οργανώσεις των ασθενών. Να δούμε τη λύπη, πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και οικονομικά με τις γραμμές των προπολογισμό για σχετικά προγράμματα δράσης. Πείτε μας λοιπόν πόσο φιλόδοξοι είσαστε. Ελπίζω να είσαστε πολύ φιλόδοξοι. Κύριε Φάγκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω κι εγώ να είμαι σύντομος για να τηρούμε και το χρονοδιάγραμμα που έχουμε. 10-15 λεπτά χρειάζομαι για να σας παρουσιάσω την ανακοίνωση της Επιτροπής και τις δυνατότητες που υπάρχουν για στήριξη των ε, οργανώσεων, όπως είπατε κι εσείς. Έρχομαι λιγάκι στη στρατηγική για την υγεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καθορίζει την προσήκησή μας ε, στον τομέα της δημόσιας υγείας. Θα ξέρετε κι εσείς και οι άλλοι ευρωβουλευτές και πυρογνώμονες ότι η κύρια ευθύνη για θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζονται σύμφωνα με τη συνθήκη ε, στα κράτη-μέλη. Είναι τα κράτη-μέλη δηλαδή που έχουν την κύρια ευθύνη για θέματα υγείας και προκειμένου για να βελτιωθεί η υγεία των ε, πολιτών. Βέβαια, συγχρόνως, εμείς έχουμε την εντολή να στηρίζουμε τα κράτη-μέλη και να προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, οικονομίες κλίμακας έτσι ώστε να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη στο ρόλο τους που είναι η βελτίωση της υγείας των πολιτών παντού στην Ευρώπη. Με την οικονομική κρίση είναι μια πρόκληση αυτή για μας και βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Γιατί θέλουμε να δούμε ότι τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να χρηματοδοτούν τις υπηρεσίες υγείας παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση τη σημερινή, αλλά θέλουμε συγχρόνως να δούμε τι θα γίνει και αργότερα λαμβάνοντας υπόψη την γύρανση του πληθυσμού, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι ο πληθυσμός της γης γυράσκει. Οι ηλικίε που οι άνθρωποι ε, παίρνουν σύνταξη, που σταματάνε να δουλεύουν, ε, αλλάζουν. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι πρέπει πράγματι να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όσο γίνεται καλύτερα τις νέες αυτές προκλήσεις. Ποιο είναι το στοιχείο κλειδί λοιπόν για τη γύρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη. Ένα από τα κεντρικά στοιχεία είναι ότι έχουμε Αλσχάιμερ και άλλες ε, ασθένειες άνοιας. Είναι λοιπόν μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο οι οικογένειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε πρόκειται για Αλσχάιμερ, είτε πρόκειται για άλλες μορφές άνοιας, το βέβαιο είναι ότι και οι πάσχοντες αλλά και όσοι ασχολούνται μαζί τους, τους φροντίζουν οι συγγενείς τους, θα υποφέρουν από αυτό. Ξέρουμε επίσης ότι πρόκειται για έναν τομέα πραγματικά δύσκολο, όχι μόνο για τις οικογένειες, αλλά και για ολόκληρο το σύστημα υγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει ανακοίνωση το 2009, είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2009, 380 τελικό κείμενο που αναφέρεται στην άνοια και το Αλσχάιμερ. Έχουμε μια στρατηγική λοιπόν η οποία βασίζεται σε τέσσερα στοιχεία κλειδί. Το πρώτο που για μας είναι πολύ σημαντικό για να στηρίσουμε τους πολίτες είναι ο πυλώνας υγεία, δηλαδή πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση. Και αυτό διότι ακόμα και αν για τις ασθένειες Αλσχάιμερ δεν έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική για την πρόληψη, για άλλες μορφές άνοιας, ιδιαίτερα αυτές που έχουν να κάνουν με την αγιακή άνοια, εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε με την πρόληψη. Δεν γνωρίζουμε πάντα αρκετά πράγματα για το τι μπορούμε να κάνουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή. Επίσης, Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε με επιτυχία να θεραπεύσουμε το Alzheimer σήμερα. Όμως υπάρχουν παρεμβάσει που βοηθούν να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα και να καθυστερήσουμε την εξέλιξη της ασθένειας. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο άμα δράσουμε στα αρχικά στάδια της ασθένειας. Βέβαια, πολύ συχνά η διάγνωση της ασθένειας έρχεται αργά. Αφού έχει περάσει η περίοδος εκείνη κατά την οποία θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα συμπτώματα. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να έχουμε καλύτερα συστήματα διάγνωσης. Οι γιατροί δηλαδή να έχουν στη διάθεσή τους τα μέσα να κάνουν έγκαιρα την διάγνωση της ασθένειας. Αυτός λοιπόν είναι ο πυλώνας υγεία που έχει να κάνει με την πρόληψη, όπως σας είπα, και με τις όσο γίνεται περισσότερες δυνατότητες ε, ε, αντιμετώπισης της ασθένειας. Έρχομαι τώρα στη δεύτερη προτεραιότητά μας. Χρειάζεται καλύτερη κατανόηση της άνοιας και όλων των μορφών άνοιας. Και αυτό είναι ζωτική σημασία για την έρευνα και τους ερευνητές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βέβαια, αντιμετωπίζουμε την άνοια σαν προτεραιότητα για μας για πολλά χρόνια τώρα. Αυτό όμως που δεν είναι πάντα γνωστό και οι συνάδελφοι στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας με ευχαριστούν πάντα που το λέω, είναι το εξή. Ή μάλλον θα σας ζητήσω να σκεφτείτε πόσοι ξέρουν το ποσοστό των κονδυλίων της έρευνας που πάνε για ευρωπαϊκό πρόγραμμα πλαίσιο. Για σκεφτείτε το. Η απάντηση είναι ότι 5% μόνο. 5% της συνολικής χρηματοδότησης. Αν θέλετε, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια τεράστια πρόκληση απέναντι μας. Πώς να αντιμετωπίσουμε το θέμα με ένα 5%. Από την άλλη μεριά, τι κάνουμε με τα άλλα 95%. Πώς μπορούμε να αποφεληθούμε και από αυτά. Γι' αυτό και μιλάμε για μια νέα πρωτοβουλία για κοινά ερευνητικά προγράμματα ώστε να μην έχουμε μόνο τις δικούς μας πόρους, αλλά να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε μαζί τα χρήματα και να καταφέρουμε να έχουμε μια καλύτερη συλλογική προσπάθεια. να έχουμε μια συνολική προσέγγιση. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να πω ότι μέχρι τώρα έχουμε επιτυχία, γιατί συμμετέχω στην πρωτοβουλία αυτή πολλές χώρες μέλη που έχουν δεσμευτεί από την πλευρά τους για αυτό τον σκοπό. Είναι μια μακροχρόνια βέβαια διαδικασία. Δείχνει όμως ότι μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο συνεργασίας. Και αυτό γιατί η πρόκληση του Αλσχάιμερ ήταν τόσο συγκεκριμένη που συμφωνήσαμε γι' αυτό. Στη συνέχεια. Ερχόμαστε στους ειδικότερου τομείς που έχουν να κάνουν με την οργάνωση των συστημάτων υγείας και τη χρηματοδότηση. Και εδώ μπαίνουμε στον πυρήνα του ζητήματος. Είπαμε πριν ότι είναι τα κράτη-μέλη που είναι υπεύθυνα για την υγεία. Όμως υπάρχουν καλές πρακτικές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν τις βρίσκουμε όμως σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, Χρησιμοποιούμε δηλαδή διάφορα μέσα προκειμένου οι βέλτιστες αυτές πρακτικές να γίνουν γνωστές και να εφαρμοστούν παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ευρωπαϊκή συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με τη θεραπεία, με την φροντίδα των πασχόντων από άνια και Αλτσχάιμερ. Και για να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, το θέμα της χρηματοδότησης της φροντίδας. Πώς χρηματοδοτείται η φροντίδα για κάποιον που έχει άνοια. Γιατί αυτή η μακροχρόνια φροντίδα και στήριξη κοστίζει πολύ. Σε πολλές χώρες μέλη, οι οικογένειές μας αντιμετωπίζουν αυτή την πρόκληση. Όταν έχεις ένα αγαπημένο σου πρόσωπο που πάσχει από άνοια Αλσχάιμερ, δεν στεναχωριούνται μόνο για την πάθηση, αλλά έχουν και οικονομικό πρόβλημα, γιατί για αυτούς για την οικογένειά τους, για την αποταμίευσή τους. Σημαίνει πολλά πράγματα μια τέτοια πάθηση. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε τον τρόπο να χρηματοδοτήσουμε τη μακροχρόνια φροντίδα για τα άτομα που πάσχουν από άνοιες. Και εδώ μπορούμε να ανταλλάξουμε ιδέες μεταξύ μας σε διάφορες χώρες. Ο τέταρτος τομέας, στον οποίο επικεντρωνόμαστε στην ανακοίνωσή μας, είναι τα δικαιώματα των πασχόντων από Άνια και Αλσχάιμερ. Σίγουρα έχουμε εδώ πέρα εμπειρογνώμονες που θα αναφερθούν σε αυτό αργότερα και που είναι πολύ πιο ειδικοί από εμά και έχουν κάνει πολύ σημαντική δουλειά σε αυτούς τους τομείς. Όμως ένα από τα σημεία που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από Άνια εξακολουθούν να είναι άνθρωποι, εξακολουθούν να έχουν τις δικές τους ανάγκες, τις δικές τους εμπειρίες και εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα να μπορούν να επικοινωνήσουν και να γίνονται σεβαστές οι επιθυμίες τους. Και αυτό πρέπει να μπει στη ζυγαριά επίσης με τη φροντίδα. Είναι δύσκολα ζητήματα αυτά. Πότε κλειδώνεις κάποιον στο δωμάτιό του από τη στιγμή που υποφέρει από άνοια. Πότε τον απομονώνεις. Και Μπορείς να μην το κάνεις, αν μπορεί, μάλλον αν δεν μπορεί να κυκλοφορήσεις ολόκληρο το σπίτι με ασφάλεια. Αυτά είναι ζητήματα που απασχολούν καθημερινά τους ανθρώπους που ασχολούνται με πάσχοντες. Γι' αυτό και χρειάζεται διάλογος για αυτά τα ζητήματα, για τα δικαιώματα, για τις ευθύνε και για την ισορροπία ανάμεσα στους διαφορούς παράγοντες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να επιβάλλει μια συγκεκριμένη προσέγγιση, θέλει όμως να προσφέρει μια πλατφόρμα διαλόγου και συζήτησης όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Τώρα για τη συγκεκριμένη στήριξη που μπορούμε να προσφέρουμε. Έχουμε χρηματοδοτήσει μια κοινή δράση υπέρ αυτών των δραστηριοτήτων υπό το πρόγραμμα Υγεία. Και χαίρομαι που μπορώ να σας πω ότι στηρίξαμε τις δύο κύριες οργανώσεις και χαίρομαι που θα τους έχουμε εδώ σήμερα αργότερα μαζί μας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις οργανώσεις αυτές και στο μέλλον. Και επίσης θέλω εδώ να τους ευχαριστήσω για την μεγάλη τους προσφορά. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σίγουρα και, άλλους, και άλλες οργανώσεις. Τέλος, κύριε Πρόεδρε. Στο μέλλον θα έχετε δει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την καινοτομία στην Ένωση. Ο πρόεδρος Μπαρόσο και οι άλλοι επίτροποι είπαν ότι θέλουμε να επικεντρωθούμε στην καινοτομία τα επόμενα χρόνια. Και σαν πειραματικό πρόγραμμα θέλουμε να δούμε την υγεία. Είναι η καινοτομία ένας από τους στόχους για το 2020. Αν δείτε λοιπόν την γύραση ε, του πληθυσμού, καταλαβαίνετε ότι η Άνια είναι άρρητα συνδεδεμένη με αυτό. Ελπίζω λοιπόν, όταν θα φτάσουμε στην εφαρμογή του, της πειραματικής αυτής πρωτοβουλίας, θα έχουμε την ευκαιρία με αυτόν τον μηχανισμό να χρηματοδοτήσουμε ακόμα περισσότερο τις ιδέες στις οποίες θα καταλήξει η σημερινή συζήτηση. Έτσι λοιπόν κύριε Πρόεδρε, μια που τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο που ξεκινούν οι νέες ιδέες, ο νέος μηχανισμός, το σημερινό εργαστήριο και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έρχονται την κατάλληλη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά όλους ιδιαίτερως την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτά τα θέματα και δεσμευόμαστε να λάβουμε υπόψη μας τα θέματα που θα συζητηθούν εδώ και στο μελλοντικό μας έργο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδοκά σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τους άλλους εμπλεκόμενους. Ελπίζουμε ότι θα ακουστούν πολύ περισσότερες ιδέες σήμερα που θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε στη δικιά μας δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank mm. Σας ευχαριστούμε κύριε Φαΐ. Ήσασταν πληρέστατος, πολύ καλή η παρουσίασή σας και βλέπουμε και την ευαισθησία που έχετε. Ε, μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιον άλλον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι ανέστητος, αλλά ε, εδώ και μήνες και χρόνια από παρουσιάσεις ήσασταν από τους καλύτερους. Ευχαριστούμε. και ελπίζω ότι όλοι όσοι συμμετέχουν σε οργανώσεις ασθενών εκτιμούν την προσήλωσή σας, την αφοσίωσή σας. Συνάδελφοι, θα περάσουμε τώρα στο επόμενο τμήμα. Θα ακούσουμε την κυρία Τσέλτον. Αλλά όχι, θα ακούσουμε την κυρία Ανερή που εκπροσωπεί την κυρία Τσέλτον. Θα θέλαμε όμως να παρακολουθήσουμε τμήματα της ταινία ε, «Το κουτί της Πανδώρας» για την οποία θα σας είχε μιλήσει η κυρία τον τώρα θα μας μιλήσει η κυρία Μαρή, ε, που βραβεύτηκε στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν του 2008 ως ε, καλύτερη ηθοποιός. Δέκα λεπτάκια θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας. Ne, zaman oldu?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 Ε, δεν ήταν ίσως και πολύ καλή ιδέα που προεδρεύω εγώ, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό, συγγνώμη. Ε, στα τουρκικά φυσικά ήταν ταινία, θα το καταλάβατε. Σαμπίνα Αγή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, εξ ονόματο τη κυρία Σέλτον, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Περιβάλλοντο και τα μέλη του σημερινού εργαστηρίου για την πρόσκληση. Δυστυχώ δεν μπόρεσε να σα θυμίσει με την παρουσία τη. Η κυρία Σέλτον επανειλημμένα συνέβαλε σε διάφορες εκδηλώσεις ε, της Λίγκας για το Αλτσχάιμερ του Βελγίου, ε, κυρίως μέσω της προβολής αυτής της ταινίας. ταινία πολύτιμη γιατί παρότι διαδραματίζεται σε άλλη χώρα, όχι στο Βέλγιο, ε, τοποθετείται στον πυρήνα του προβλήματος γιατί καταδεικνύει όλες τις ε, αλλαγές που σημειώνονται μέσα στην οικογένεια με την εμφάνιση της νόσου. Η νόσος ε, του Αλτσχάιμερ δεν είναι κάτι ορατό απαραίτητα ε, αλλά η πουλά εγκαθίσταται σε, στην οικογένεια και όλοι πρέπει να επανατοποθετηθούν αντιμέτωποι με, με άγνωστη κατάσταση, ε, με γεγονότα που εκπλήσουν, που δεν κατανοούμε απαραίτητα, γιατί δεν γίνεται εκούσια αυτό, υφίσταται κάποιος την νόσο, όπως και η οικοί του εξάλλου. Αυτό δείχνει ότι αγωνίζεται η οικογένεια και για να βρει λύσεις ε, για τον ασθενή, αλλά και για τους ίδιους. Ρώτησα λοιπόν ε, την κυρία Σέλτον ε, γιατί πραγματικά διαδραματι... έπαιξε με εξαιρετικό τρόπο το ρόλο της ασθενούς αν έχει διαβουλευτεί με κάποιους που γνωρίζουν την όσο και μου είπε όχι, εγώ είμαι ηθοποιός, ε, μου απέδωσαν αυτό το ρόλο ε, και ε, αυτό που έκανα είναι ότι μιμήθηκα. Αυτό αυτούς τους ανθρώπους ε, και αυτή είναι η απόδειξη του ταλέντου της. Ε, σας προσκαλώ δεν να δείτε ολόκληρη την ταινία γιατί πραγματικά χρησιμοποίησε όλα τα μέσα που είχε στη διάθεσή της, όλες τις σκηνές, όλες τις συμπεριφορές ε, για να περιγράψει τις δυσκολίες που συνεπάγεται αυτή η νόσος. Από τι οφόρο τιμής και πάλι σε αυτήν την ηθοποιό τόσο αυθεντική, τόσο ταλαντούχα η κυρία Σέλτον είναι 99, χρονών ε, και η καταπληκτική της παρουσία μέσα σε αυτή την ταινία αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα για μια καλή γύρανση. Όσοι χάνουν αυτή την γνωσιακή λειτουργία και δεν μπορούν πλέον να εκφραστούν, ε, αξίζουν παρόλα αυτά μια ε, ποιοτική γύρανση. Δεν μπορούμε να τους τιμωρήσουμε διότι νοσούν ε, και πρέπει να τους υποστηρίξουμε, πρέπει να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση και χαίρομαι εκ των προτέρων για τη διεξαγωγή του σημερινού εργαστηρίου. Ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστούμε πολύ τη Σαμπίν Άρη. Και συνεχίζουμε τώρα στο πρώτο τμήμα. Ε, μάλλον τελείωσε πρώτο πρέπει στο δεύτερο τμήμα που είναι οι εμπειρογνώμονε μας και εκπρόσωποι των ασθενών. Αυτοί που στη δουλειά τους, στην καθημερινή του ζωή βρίσκονται μαζί με τους πάσχοντες. Θα μας πούνε τη γνώμη τους, πώς πιστεύουν ότι πρέπει να χειριστούμε το Αλσχάιμερ και την άνοια. Θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στον Ζαν Ζορς που είναι ο διευθυντής της Alzheimer Europe. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλείτε να έρθω στη σημερινή σας συνεδρίαση. Ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βλέπω εδώ διάφορους συναδέλφους και φίλους μάλιστα που συμμετέχουν στην οργάνωσή μας και μας στηρίζουν για μας και τις εκστρατείες μας. Για μένα αυτού του είδους η συνεδρίαση είναι η ολοκλήρωση της εκστρατείας μας. Δηλαδή έτσι αναγνωρίζουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τη δουλειά μας. Απ' την άλλη μεριά αποτελεί και ένα νέο σημείο κίνησης για την συνέχεια του έργου μας. Ελπίζω και εγώ πως ε, θα προσφέρουμε σήμερα κάτι παραπάνω για την ε, καταπολέμηση της άνοιας και για την βελτίωση των συνθηκών ζωής των πασχόντων. Πολύ συχνά ερχόμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε ότι τα ευρωπαϊκά κοινοτικά όργανα δεν κάνουν αρκετά πράγματα. Ε, λοιπόν, για μια φορά έχουμε έρθει εδώ για να ευχαριστήσουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τη δουλειά που κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν στο μέλλον. Ναι. Θέλω να μιλήσω λοιπόν εκ μέρους της οργάνωσής μου. Έχουμε 31 ενώσεις που συμμετέχουν από 28 χώρες. Αυτό που θέλω πάνω απ' όλα σήμερα να σας πω είναι κάποια στοιχεία. Όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και εμείς βάζουμε σαν προτεραιότητα το Alzheimer. Πρέπει να ξέρουμε ότι ένα από τα στοιχεία κλειδί, η ενημέρωση που θέλει ο κόσμος δηλαδή, είναι ότι πόσοι υποφέρουν από την ασθένεια αυτή. Χάρη λοιπόν στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορέσαμε να κάνουμε μια έρευνα για τρία χρόνια όπου αναλύσαμε τα περιστατικά που έχουμε. Η ομάδα των ερευνητών μας είπε ότι έχουμε 194 άρθρα, από τα οποία 74 αναφέρονται στα κριτήρια ποιότητας που έχουν αναπτυχθεί από διάφορες επιστημονικές ομάδες. Προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε ποια είναι η κατάσταση ανελικία, αν υπάρχει διαφορά δηλαδή ανάμεσα στη δικιά μας τη δουλειά και την ε, δουλειά που έχει γίνει παλιότερα, δεκαετία του 90 από το Γιούροντα. Στη διαφάνεια αυτή λοιπόν για τους άντρες βλέπετε ότι υπάρχει μικρή διαφορά ανάμεσα σε αυτά που βρήκαμε εμείς και σε αυτά που βρήκε η Eurodem. Τώρα κατά πόσο υπάρχει μεγάλη διαφορά ή όχι διαφορά, αν υπάρχει, υπάρχει όσον αφορά τον επιπολασμό στις γυναίκες. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 υπήρχε διαφορά σε μεγάλες ηλικίε. Γιατί εμείς βρήκαμε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση σύμφωνα με την ηλικία. Δηλαδή από μια ηλικία και μετά οι γυναίκες υποφέρουν πολύ περισσότερο. Μία στις δύο γυναίκες κινδυνεύει να αντιμετωπίσει νοητικά προβλήματα κάποια στιγμή. Κάναμε λοιπόν υπολογισμούς για να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία ε, για να δούμε πόσοι άνθρωποι υποφέρουν από Αλσχάιμερ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι διαπιστώσαμε. Εδώ υπάρχει κάποιο λάθος από τη δικιά μου την πλευρά. είναι 7,4, είναι 7,3 εκατομμύρια. 7,3 εκατομμύρια άνθρωποι λοιπόν στην Ευρώπη έχουν ε, άνοια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διπλασιαστεί και θα τριπλασιαστεί το νούμερο αυτό μέχρι το 2050. Και εδώ το παγόβουνο που βλέπετε δεν είναι μόνο για να σας δείξουμε ότι τα νούμερα που έχουμε σήμερα είναι πολύ λιγότερα από αυτά που θα έχουμε στο μέλλον, αλλά επειδή και από το έργο αλλά και από τις ερευνές μας βρήκαμε ότι άνθρωποι οι οποίοι ε, έχουν διαγνωστεί ανοικοί πολύ συχνά είναι πολύ λιγότεροι ε, από αυτούς που επηρεάζονται από την ασθένεια, διότι υπάρχουν οι συγγενείς τους, τα παιδιά τους, αυτοί που τους φροντίζουν. Η κυρία Βασιλείου, η Επίτροπος για την Υγεία, έχει μιλήσει για 90 εκατομμύρια Ευρωπαίους που επηρεάζονται από την ασθένεια, αν δηλαδή δεν λάβουμε υπόψη μας μόνο τους πάσχοντες, αλλά και τους συγγενείς τους και τους ανθρώπους που τους φροντίζουν. Κοιτάξαμε επίσης τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα όσους εκπονούν πολιτική. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα για αυτά γιατί δεν έχω αρκετό χρόνο, αλλά πρέπει να σας πω ότι ο υπολογισμό για το κόστος ε, της ε, άνοιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση του, τον 27 το 2008 ήταν 160 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 56% ήταν για άτυπη φροντίδα. και αν δούμε το συνολικό κόστος ευρύτερα, είναι 167 εκατομμύρια. Τι, δισεκατομμύρια, συγγνώμη. Τι σας, ε, τι εννοώ αυτά και το βλέπετε αυτό σε αυτήν την ε, εικόνα. Δείτε αναχώρα. Συμφωνούμε με τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η άνοια αποτελεί προτεραιότητα αλλά συμφωνούμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την έγκαιρη διάγνωση και τα δικαιώματα των πασχόντων. Όταν φτάνουμε λοιπόν στο θέμα της διάγνωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να βελτιώσει, είπε, την έγκαιρη διάγνωση σε αρχικό στάδιο. Εμείς ρωτήσαμε τους ανθρώπους που φροντίζουν τα άτομα με τις πόσο καιρό σας παίρνει ε, μέχρι να ανακαλύψετε ότι υπάρχουν ε, τέτοια κρούσματα, ότι οι άνθρωποι με τους οποίους δουλεύετε τελικά έχουν Αλσχάιμερ ή κάποια άλλη μορφή άνοιας. Και να, στη Γερμανία έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Σε 10 μήνες. Χρειάστηκαν δηλαδή 10 μήνες από τη στιγμή που κάποιος ασχολείται με τη μητέρα του, με τον πατέρα του, ένα συγγενή του τέλο πάντων, του χρειάστηκαν 10 μήνε για να καταφέρει να φτάσει στη διάγνωση ότι πάσχει από κάποια μορφή σε άλλε χώρε του παίρνει πολύ περισσότερο καιρό. Σε χώρε όπω είναι η Γαλλία του παίρνει δύο χρόνια και στο Ηνωμένο Βασίλειο 32 μήνε. Τουλάχιστον έτσι μα είπαν ότι του χρειάστηκαν 32 μήνε για να καταλάβουν ότι κάτι δεν. από τη στιγμή που κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά, μέχρι να έχουν τη διάγνωση για την ασθένεια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει μεγάλε επιπτώσει. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θέλει ανταλλαγή πληροφοριών για τι πρακτικέ φροντίδα. Έχουν γίνει κάποιες έρευνες από την Alzheimer Europe το 2006 που ρώτησε τους περιθάλπτοδες πόσος χρόνος τους χρειάζεται ε, για να ασχολούνται με τον ασθενή. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο αρχικό στάδιο και το πιο προχωρημένο στάδιο βέβαια. 20% για ένα στου τέσσερι περιθάλποντε είπε ότι τουλάχιστον 10 ώρες την ημέρα ασχολείται με το άτομο που έχει άνοια. Και όταν λέμε φροντίδα, εννοούμε ότι πρέπει να είσαι στον ίδιο χώρο, στο ίδιο δωμάτιο, για να ξέρει ότι ο ασθενής δεν θα κάνει κακό στον εαυτό του, δεν θα χτυπήσει. Δεν μιλάμε για εντατική φροντίδα, αλλά εννοούμε ότι πρέπει να είσαι εκεί, να βρίσκεσαι στο ίδιο δωμάτιο με τον ασθενή. 39% φτάνει σε ένα μεσαίο στάδιο που μας λένε ότι θέλουν 23% ε, του χρόνου και 50% μας λένε ότι θέλουν πάνω από 10 ώρες την ημέρα να βρίσκονται με τον ασθενή. Στην ίδια μελέτη ρωτήσαμε και τους περιθάλπτοντες να μας μιλήσουν για τις υπηρεσίες που πιστεύουμε εμείς ότι είναι ζωτικές σημασίες για αυτούς, για να μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς. Εδώ δεν θα σας αναφέρω ολόκληρη την μελέτη, αλλά τι λένε. Αυτοί που λένε ότι 10 ώρες τουλάχιστον ασχολούνται με τους ε, ασθενείς, λένε ότι χρειάζονται παραπάνω βοήθεια. Ένας στους τρεις λένε ότι χρειάζονται respite care για τους ασθενείς αυτούς. Η Γερμανία είπε 51% από τους περιθάλποδες ότι θέλουν εξασφάλιση προσωρινής μέρημνας εκτός κατοικίας, να μεταφερθούν δηλαδή κάπου αλλού οι ασθενείς. Στην Ισπανία μόνο 3% των ανθρώπων που ασχολούνται με ασθενεί είπαν ότι θα του βοηθούσε αν πήγαινε ο ασθενής εκτός σπιτιού. Προτιμών να έρχεται κάποιο στο σπίτι ή να πηγαίνουν μαζί με τον ασθενή κάπου κατά τη διάρκεια της ημέρας για να μπορούν να έχουν λίγο χρόνο να πάνε στο κομμωτήριο, να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους, αντί να είναι συνέχεια με τον ασθενή. Αλλά μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όχι συνολικά. Το θέμα των δικαιωμάτων τώρα, το θέμα της ηθικής. Ρωτήσαμε επίσης τους περιθάλποντες, ο ασθενής με τον οποίο ασχολείστε ξέρει ότι έχει άνοια ή Αλσχάιμερ. Εδώ βλέπετε το μέσο όρο 65% είναι ο μέσος όρος, αλλά υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Στη σκοτή 80% είπαν ότι ναι, το ξέρουν οι ασθενείς ότι έχουν άνοια η Αλσχάιμερ αλλά μόνο 23% στην Ισπανία. Άρα λοιπόν όταν μιλάμε για ανταλλαγή των πρακτικών όσον αφορά την ηθική, όπως ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θέλεις να έχει το άτομο μεγαλύτερη αυτονομία, αν θέλουμε να τους Θέλουμε πλήρης ανθρώπου, το βασικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν τι έχουν. Και έτσι να συμμετέχουν και αυτοί σε ό,τι αποφάσεις λαμβάνονται που τους αφορούν σε κάποιο στάδιο της ζωής τους, ώστε να μπορούν να προλάβουν τη συνέχεια ή να φροντίσουν για το μέλλον τους. Το 2006 η οργάνωσή μας κατέληξε στη δήλωση των Παρισίων. Εκεί ορίσαμε προτερότητες στο θέμα της δημόσιας υγείας, της ιατρικής και των προτεραιοτήτων των επιστημονικών, για τη φροντίδα, για την ηθική και τα νομικά ζητήματα και για τις ε, οργανώσει Αλσχάιμερ. Αυτό το οποίο θέλουμε και αυτό που ζητάμε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι να, να αναγνωρίσουν την άνοια σαν προτερότητα σε θέματα δημόσιας υγείας. Θέλουμε επίσης περισσότερα εθνικά προγράμματα δράσης. Θέλουμε και καλύτερο συντονισμό στην Ευρώπη για την πρόληψη και την θεραπεία. Τέλος θέλουμε περισσότερα κονδύλια για την έρευνα όσον αφορά την άνοια και το Alzheimer. Αυτές είναι οι προτεραιότητες κλειδί που έχουμε εμείς και που ζητάμε να υιοθετήσουν και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν θα σας εκπλήξει να ακούσετε ότι εφόσον εμείς εκπροσωπούμε πάσχοντες και περιθάλπτοντες, εννοείται ότι στηρίζουμε απόλυτα ό,τι πρωτοβουλίες λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ αυτών. Θέλουμε, όπως σας είπε, εθνικά προγράμματα πλαίσιο. Και είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Είπε και ο ότι η Επιτροπή χρηματοδοτεί τη συνεργασία και τον συντονισμό των προσπαθειών που γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται συντονισμό και συνεργασία και με την κοινωνία των πολιτών, με τις οργανώσεις δηλαδή των πασχόντων από Άνια. Και αυτό είναι κάτι που κοστίζει. Και αυτό είναι που κάνουμε εμείς για να στηρίξουμε τους πάσχοντες και αυτούς που τους φροντίζουν. Θέλουμε να αναγνωριστεί αυτή η δουλειά και να χρηματοδοτηθεί και αυτή στο μέλλον. Πάντως εσείς που καθορίζετε την πολιτική. Ένα τελευταίο μήνυμα. Πώς πρέπει να δράσουμε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Συνεργασία μεταξύ των ε, κρατών μελών για τα θέματα πασχόντων και περιθάλπτοντων και το πρόγραμμα δημόσιας υγείας που θα επαναξεταστεί σύντομα να λάβει υπόψη αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει η Άνια και το Αλσχάιμερ να έχουν ακόμα μεγαλύτερη προτεραιότητα. Μέχρι τώρα έχουμε πετύχει την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί θα στηρίξετε την εκκλησία μας και θα δώσετε μεγαλύτερη θέση στα προγράμματά σας για την Άνια και το Αλσχάιμερ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω σας άξεγαν τα συγχαρητήρια και προτείνω να συνεχίσουμε γιατί έχουμε καθυστερήσει λιγάκι και πρέπει να μείνει λίγος χρόνος για συζήτηση. Θα ήθελα να σας συστήσω τον κύριο Φασόνη, ο οποίος ε, είναι αναπληρωτής επιστημονικός διευθυντής ε, του Εθνικού Κέντρου ε, Έρευνας Alzheimer Disease, ασθένεια Alzheimer στην Ιταλία. Και ο κύριος Φριζόνη, χρειάζεται το λάπτοπ του, κάποιο λάπτοπ, κάποιον υπολογιστή φορητό, για να μπορεί να κάνει την παρουσία του. Ε, μπορούμε λοιπόν με μεγάλη μας ε, χαρά να ακούσουμε την επιστημονική προσέγγιση και την ερευνητική του κυρίου Φριζόνη. Thank you, Mrs. Vice President. Uh, Honorable Matthias, thank you for this Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ε, Πρόεδρε και αγαπητά μέλη της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, και του Κοινοβουλίου για την πρόσκληση που μας απευθύνατε. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω την προοπτική ενός ευρωπαϊκού κλινικού επιστήμονα για το Alzheimer εγώ ε, και δέχομαι ασθενείς και κάνω έρευνες στην ασθένειά τους. Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι αυτά τα οποία θα σας πω ε, θα αντιστοιχούν πλήρως με αυτά που θα σας πούνε και άλλοι ερευνητές στην Ευρώπη, αλλά θεωρώ ότι αυτά τα οποία θα σας πω εγώ ε, τα συμμερίζονται αρκετοί επιστήμονες στην Ευρώπη.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 Λοιπόν, ε, θα ήθελα να ασχοληθώ με ορισμένα θέματα. Θα ήθελα να δαπανίσω λίγο από το χρόνο σας για να σας ενημερώσω για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά στην παθοφυσιολογία της ε, νόσου Αλτσχάιμερ. Δεν είναι όλες οι μορφές άνοιας Αλτσχάιμερ, όπως και όλες οι μορφές καρκίνου, δεν είναι καρκίνος του πνεύμονα. Η ασθένεια Αλτσχάιμερ είναι η πιο συνηθισμένη. Και τώρα αρχίζουμε ε, να μπορούμε να εικάσουμε ε, γιατί προκύπτει αυτή η ασθένεια. Έχουμε κάποιες καλές ενδείξεις. Η παθοφυσιολογία και η έρευνα στην παθοφυσιολογία μπορεί να βοηθήσει τους ε, ασθενείς. Ε, και αυτό γίνεται τώρα, ακριβώς αυτή τη χρονική περίοδο. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας παρουσιάσω ε, την έρευνα στην νόσο Alzheimer στην Ευρώπη και αυτό από κλινική σκοπιά. Και θα ήθελα να ασχοληθώ με την έρευνα, όπως επίσης ε, και με το θέμα της ε, ανακάλυψης νέων γνώσεων. Να δούμε λοιπόν γιατί προκύπτει η ασθένεια Alzheimer. Στον εγκέφαλο σωρεύονται τοξικές πρωτεΐνες οι οποίες ε, βιταμιλοειδή και αυτές σωρεύονται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Για πολλά χρόνια, 20 άλλοι είναι 30 χρόνια, αυτή, αυτή η απόθεση τοξικών ουσιών στον εγκέφαλο δεν φαίνεται, δεν, δεν παρουσιάζονται συμπτώματα. Και σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία ας υποθέσουμε στα 75 σε έναν ε, ε, εικονικό ασθενή ε, εμφανίζονται πολύ ήπια συμπτώματα ε, ξεχνάει κανείς πράγματα κάτι που παρουσιάζεται σε πολλούς από εμά ξεχάσαμε τα κλειδιά μας ξεχάσαμε που έχουμε παρκάρει το αυτοκίνητό μας τέτοιου είδους ενδείξεις όμως καμία αναπηρία οι άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά, φυσιολογικά και μέχρι πριν από λίγα χρόνια προέκυψε από τη σώρευση αυτών των τοξικών ουσιών άνοια. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι πλέον δεν μπορούσαν να εργαστούν, είχαν αναπηρία. Δεν μπορούσαν να συνεχίσουν την κανονική του ζωή. Η άνοια λοιπόν, αυτό γνωρίζαμε μέχρι τώρα. ο Ζαν Ζόρζ με αυτό ακριβώς ασχολήθηκε. Με την άνοια. Και από τη στιγμή ε, που εμφανίζονται τα συμπτώματα μέχρι τη διάγνωση, αυτή είναι η άνοια και η... στον εγκέφαλο όμως η ε, νευροβιολογική κατάσταση είναι πολύ πιο παλαιότερη. Βλέπετε λοιπόν ότι διαδίδεται η νευροπαθολογία και στον εγκέφαλο μπορούμε να διαπιστώσουμε την νευροπαθολογία στον εγκέφαλο και την φάση της άνοιας. Ε, ο εγκέφαλος είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος. Σε αυτή λοιπόν τη φάση Ακριβώς σε αυτή τη φάση, παραδοσιακά, ε, μέχρι τώρα τουλάχιστον, κάναμε τη διάγνωση της νόσου Alzheimer με βάση κλινικά κριτήρια. Ε, δεν χρειαζόμασταν ιδιαίτερα εξελιγμένες ε, και ταπανηρές μεθόδους. Ε, στα συμπτώματα, κυρίως όσον αφορά στη μνήμη, δεν υπήρχε αναπηρία. Ο εγκέφαλος είναι αρκετά επιβερημένος με τοξικές πρωτεΐνες, προφανώς, ε, ο εγκέφαλος έχει μια νευρολογική, νευροβιολογική, ε, ένα νευροβιολογικό ιστορικό εναπόθεση τοξικών ουσιών. Και σε αυτή τη φάση τώρα πιστεύουμε πλέον ότι μπορούμε να διαγνώσουμε την νόσο. Με αυτό μπορούμε να το πράξουμε με ε, βιολογικούς δείκτες και με τις απεικονίσεις, την απεικονιστική. Βέβαια, ακόμα δεν μπορούμε να διαγνώσουμε την ασθένεια στη φάση όπου εμφανίζονται όλα τα συμπτώματα, αλλά εκεί θέλουμε να βαδίσουμε. Ας δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι διαγνωστικοί δείκτες. Ένας εξ αυτών είναι η ατροφία. Η ατροφία του υποκάμπιου, που είναι ε, μια μικρή δομή ως ένα μικρό δαχτυλάκι ε, που είναι βαθιά ενταγμένο στον εγκέφαλο μπορεί κανείς να εντοπίσει την αυτροφία. Πολλοί νευρώνες ε, μπορούν ε, να μεταφέρουν μηνύματα απεικόνηση μαγνητικού συντονισμού και ο δεύτερος ε, δείκτης είναι ο μεταβολισμός. Υπάρχουν ε, κάποιοι ε, τομείς που δεν μπορούν πλέον να καταναλώσουν τη γλυκόζη. Μπορούμε να εντοπίσουμε αυτή την, το σύμπτωμα. Και το τρίτο είναι ότι μπορούμε να πάρουμε ένα δείγμα από τον νοτιέο μυελό και από εκεί να κάνουμε ακριβείς μετρήσεις. Οι ασθενείς με Alzheimer παρουσιάζουν κάποιο συσχετισμό αυτών των δύο πρωτεϊνών. Και το τελευταίο παράδειγμα είναι, όπως ε, σας είπα, τα αμυλοειδή Εκεί κάνουμε μια τομογραφία νευρώνων. Είναι η νέα τεχνική, η οποία είναι μια κλινική πραγματικότητα ε, και θα είναι μάλλον κλινική πραγματικότητα ε, περίπου σε 18 μήνες από τώρα. Έτσι λοιπόν θα αλλάξει ριζικά εικόνα για το πώς ε, διαγνώσκεται η ασθένεια. Γιατί πρέπει να γίνεται πιο έγκαιρα διάγνωση, διότι επιθυμούμε να εντοπίσουμε την ασθένεια το συντομότερο δυνατόν και το συντομότερο δυνατόν σημαίνει όταν εμφανίζονται τα ήπια συμπτώματα ε, απώλειας ή ανεπάρκειας της μνήμης. Να εντοπίσουμε λοιπόν τα πρώτα συμπτώματα, να χορηγήσουμε φάρμακα τα οποία θα διακόψουν ή τουλάχιστον θα επιβραδύνουν την ε, εναπόθεση ε, των πεπτιδίων αμυλοειδούς β και να μπορέσουμε να καταστήσουμε πιο ήπια την καμπύλη έτσι ώστε ο ασθενής να παραμείνει σε ήπιες διαταραχές μνήμης χωρίς αναπηρία το οποίο βέβαια σημαίνει για τον ίδιο υψηλή ποιότητα ζωής. Εσείς θα μπορούσε να πει «Μα όλα αυτά είναι επιστημονική φαντασία» κάθε άλλο. Ήδη τώρα γνωρίζουμε ότι μπορούμε να καθαρίσουμε τον εγκέφαλο από τα πεπτίμια αμυλοειδούς β' Έχουμε κάνει μια κλινική μελέτη με αντισώματα και αυτό που βλέπετε εδώ είναι πεπτίδια αμυλοειδούς β στον ασθενή πριν και μετά την αγωγή με αυτά τα φάρμακα και βλέπουμε, είναι προφανές, ότι μειώνται σημαντικά τα αμυλοειδή β μετά την ε, αγωγή. Και αυτά, αυτή η θεραπεία γίνεται με εικονικά φάρκα, πλασίμπο και όχι πραγματικά δραστικά φάρμακα. Μπορούμε λοιπόν να αφαιρέσουμε τα αμυλοειδή β από τον εγκέφαλο. Δυστυχώς αυτή οι ασθενείς, παρότι αφαιρέσαμε τα αμυλοειδή, δυστυχώς επαναλαμβάνω, στην κλινική του εικόνα παρουσιάζουν συνέχιση της ασθένειας, της νόσου. Ε, είμαστε στη φάση όπου μπορούμε να αφαιρέσουμε τα αμυλοειδή β, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να ε, αναχαιτήσουμε τον περαιτέρω εκφυλισμό. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Υπάρχει μια σειρά φαρμάκων για την... Ε, βρίσκονται τα φάρμακα στη φάση των κλινικών δοκιμών και αυτά θα μπορέσουν να τροποποιήσουν την εξέλιξη της νόσου. Και αν είναι δραστικά, ενδέχεται κατά τα επόμενα έτη να εμφανιστούν στην αγορά, αν αποδειχθούν δραστικά. Ως ερευνητέ τώρα, πώς μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες. Πώς συγκεντρώσαμε αυτή τη γνώση. Υπάρχει ένα καθοριστικό στοιχείο που ήταν οι μεγάλες οριζόντιες ε, πολυκλαδικές μελέτες σε πολλούς τομείς που σημαίνει ότι πήραμε μεγάλο αριθμό ασθενών με καθόλου ή και με ήπια συμπτώματα ε, κάναμε σκάνινγκ CSF πήραμε τους πιο σημαντικούς δείκτες και τους παρακολουθήσαμε μέσα στη διάρκεια του χρόνου από δύο μέχρι πέντε χρόνια όσο μπορέσαμε, όσο ήταν δυνατό και εφικτό. Κάναμε λοιπόν μια μεγάλη σειρά πολυκλαδικών μελετών και όπως μπορείτε να φανταστείτε οι μελέτες αυτές είναι αρκετά δαπανηρές. Ας δούμε που βρίσκεται η Ευρώπη σήμερα όσον αφορά την όσο. Αυτές ε, οι οριζόντιες ε, μελέτες και υπάρχει ένας ε, μεγάλος αριθμός εξ αυτών ε, που χρηματοδοτήθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως βλέπετε εδώ, η μεγαλύτερη έλαβε χώρα στις Ηνωμένε Πολιτείε, ADNI, είναι μια πρωτοβουλία που έγινε για το Alzheimer. Παρεμφερή έρευνα έγινε και στην Αυστραλία και στην Ευρώπη έλαβε χώρα μία μελέτη, μικρότερη βέβαια, αυτή έλαβε χώρα το 2007 και τώρα έχουμε μία καινοτόμα μελέτη η οποία ε, συνεχίζει να τρέχει. Και στην Ιαπωνία ε, έχουν χρηματοδοτηθεί παρεμφερείς μελέτες. Η Ευρώπη λοιπόν είναι ένας ε, από τους χώρους που δραστηριοποιείται σε αυτό το θέμα. Η συγκέντρωση των δεδομένων και μιλάμε για μεγάλες ε, και έντονα οριζόντιες μελέτες οι οποίες μας επιτρέπουν τη συγκέντρωση δεδομένων. Βέβαια, ε, το να συγκεντρώνει κανείς τα δεδομένα, καλό είναι αυτό. Από την άλλη όμως, το να αποκομίσει κανείς γνώση από τα δεδομένα, αυτό είναι η δεύτερη φάση για να μπορέσει κανείς να ε, καθορίσει τους ε, δείκτες διάγνωσης, ε, εξέλιξης και να κατανοήσει κανείς καλύτερα την παθοφυσιολογία της νόσου. Για να μπορέσουμε λοιπόν να αποκομίσουμε γνώση από τα δεδομένα χρειαζόμαστε την απαραίτητη επιστημονική υποδομή. Χρειαζόμαστε χώρους αποθήκευσης αυτού του τεράστιου όγκου των δεδομένων και χρειαζόμαστε και τα εργαλεία για να μπορέσουμε να αποκομίσουμε ε, πληροφορία από την απεικόνηση, κάτι που δεν είναι τόσο απλό. Και τέλος, αυτή τη γνώση πρέπει να τη μεταφέρουμε σε κλινική πρακτική, σε κάτι που να είναι χρήσιμο για τον ε, πάσχοντα. Ακριβώς λοιπόν όταν πρόκειται για τη μεταφορά αυτής της γνώσης σε κάτι που να είναι χρήσιμο για τον Πάσχοντα, εκεί παίζει ρόλο η τυποποίηση, η ε, ανάπτυξη διαδικασιών έτσι ώστε ε, να μπορεί να γίνει ανάγνωση των διαγνωστικών ε, δικτών. Γιατί να μπορούμε να διαγνώσουμε το διαβήτη ή τον καρκίνο του προστάτη διότι μπορούμε να μετρήσουμε τη γλυκόζη στο αίμα και μπορούμε αυτό να το κάνουμε στην Ιταλία, στην Πολωνία, οπουδήποτε. Η γλυκαιμία η δική μου θα είναι 95% οπουδήποτε και αν τη μετρήσουμε. Αυτό είναι κάτι ε, που πρέπει επίσης να το επιτύχουμε με τους ε, διαγνωστικούς ε, δείκτες για την νόσο Αλτσχάιμερ. Αυτές τουλάχιστον είναι οι προσπάθειες των Ευρωπαίων επιστημόνων. Αυτό ε, καλό είναι. Βέβαια χρηματοδοτείται αυτή η έρευνα από την Αμερικανική Ένωση Αλτσχάιμερ. Καλό και αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ίσως ε, θα έπρεπε μερικοί να το σκεφτούν κάποιοι, ίσως ε, θύνονται στην Ευρώπη. η Ευρώπη εμπλέκεται ιδιαίτερα στο να προσφέρει την υποδομή στους επιστήμονες. Ε, καταβάλλονται τουλάχιστον ε, δύο ειδών προσπάθειες που αποσκοπούν στο να υπάρξει ένα παγκόσμιο εργαστήριο απεικονιστικής. Αυτό το χρειάζονται οι επιστήμονες όπως σας είπα, για να μπορούν να αποκομίσουν γνώση και πληροφορίες από τις ε, εικόνες ε, ε, από τις διάφορες απεικονιστικές διεργασίες και εκείνο που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που γι' αυτό μας χρηματοδοτηθεί, είναι για να μπορούμε να φτιάξουμε ένα παγκόσμιο εργαστήριο απεικονιστικής, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα εναρμόνισης. Δηλαδή, υποδομές που υπάρχουν ε, σε διάφορα εργαστήρια να είναι συμβατές με υποδομές που υπάρχουν ε, στην Βόρεια Αμερική, της Ευρώπης ας πούμε, με αυτές της ε, Βόρειας Αμερικής. Και εδώ η Ευρώπη διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Για να ολοκληρώσω, όπως βλέπετε και μόνοι σας, τα τελευταία 20 χρόνια η έρευνα του νόσο Αλσχάιμερ έχει κάνει μεγάλα άλματα, έχει κάνει άλματα ως προς την πρόοδό της και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε ε, βάσιμες ελπίδες για διάγνωση και ε, στο εγγύς μέλλον και ε, να, για φάρμακα τα οποία θα επηρεάζουν την εξέλιξη της νόσου. Στην Ευρώπη συγκεντρώνονται γνώσεις ε, και αναπτύσσονται ε, και υπηρεσίες ε, που προσφέρονται στην επιστήμη. Οι επιστήμονες βέβαια ίσως πρέπει να αναπροσαρμοστούν έτσι ώστε και οι Ευρωπαίοι επιστήμονες να χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς φορείς. Και η κλινική έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι αναπτύσσονται πολυκλαδικές ε, εξελιγμένες μελέτες που αυτές όμως χρειάζονται περισσότερα κίνητρα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Dr. Fessoni, thank you very much. Dr. Fessoni, ευχαριστούμε πάρα πολύ. That was for, for all of us very interesting for some... Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση ε, για όσους δεν γνωρίζουν ενδελεχώς το ζήτημα, αλλά μας δώσατε πολύ καλές ιδέες. Και όπως είπε και ο κύριος Φαγή και ο κύριος Ζόλς, ε, χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία. Ε, τώρα θα ακούσουμε την κυρία Καπούτο από την Διεθνή Ψυχοαναλυτική Ομοσπονδία. Παρακαλώ. Prima di iniziare la mia Πριν ξεκινήσω θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστώ τη Μαρίζα Ματίες γιατί μου προσέφερε τη δυνατότητα να βρίσκομαι εδώ και να ακούσω ε, πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρεμβάσεις. Ε, υπάρχουν ε, δύο άτομα δικά μου, πολύ γνωστά, οικία, που ε, νόσησαν και πέθαναν από την νόσο Αλτσχάιμερ. Έτσι λοιπόν ε, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ε, το τι ακριβώς διαδραματίστηκε, τα βιώματα των οικείων με αυτή την ασθένεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαρίζα και για ένα άλλο λόγο, διαφορετικό, επαγγελματικό, διότι η δραστηριότητα του ψυχοαναλυτή ε, κατά κανόνα ε, συνδυάζεται ε, με την πολυθρόνα, το κρεβάτι, ίσως και μια πίπα που καπνίζει ο ψυχαναλυτής και υπάρχει αυτή η εικόνα διεθνώς ότι ο ψυχαναλυτής είναι κλεισμένος σε μία αίθουσα και δεν συνεργάζεται με ερευνητικές δραστηριότητες όχι μόνο όσον αφορά την ψυχιατρική αντιμετώπιση της νόσου αλλά και την κλινική. γιατί έχουμε καταρχήν την ε, δυστροφία, την μυϊκή δυστροφία και αυτή μπορεί να καταλήξει ε, τελικά σε Alzheimer. Ως εκ τούτου η δουλειά του ψυχαναλυτή είναι πολύ σημαντική. Είναι σημαντικό να συνεργάζεται μέσα σε μία ομάδα. Είναι σημαντικό να συνεργάζεται βέβαια και με τους οικείους ε, του Πάσχοντας και με τον ίδιο τον Πάσχοντα. Η δική μου λοιπόν η παρέμβαση έχει ως ε, αντικείμενο ε, τον χώρο της ε, απώλειας μνήμης. Υπάρχουν ενδείξεις που όμως από τις οποίες μπορεί κανείς να καταλήξει μόνο στο ότι υπάρχει απώλεια της μνήμης. Και ε, γνωρίζω ότι εδώ υπάρχουν ε, δύο διαφορετικές λειτουργίες που είναι συνδεμένες μεταξύ τους, η συνειδητή και η ασυνείδητη φάση και που μπορεί κανείς να τις εξηγήσει αυτές τις ε, δύο φάσεις. Ο χρόνος βρίσκεται σε άμεση σχέση με την λειτουργία του εγκεφάλου. Ο χρόνος της ασυνειδησίας μπορεί όμως να συμπέσει και με το χρόνο της συνείδησης. Ως εκ τούτου προκύπτει μια διαλεκτική ανάμεσα στην μνήμη και την απώλεια μνήμης. Ε, εδώ δεν μιλάμε για μια προσωρινή ασθένεια είναι ότι χάνει κανείς τη συνείδηση αυτών που έχει βιώσει και έχει ζήσει. Ε, είναι περίεργα τα παιχνίδια που παίζει η μνήμη. Σιγά σιγά ε, χάνεται η μνήμη, ε, προκύπτει η απώλεια. Ως εκ τούτου ε, κάποιος που έχει συνειδητές και ασυνείδητες μνήμες, ο άνθρωπος αυτός συνεχίζει να ζει. Ήδη ο Πλάτωνας είχε μιλήσει για την απώλεια μνήμης και είχε πει ότι μπορεί να συγκαλυφθεί, δεν μπορεί όμως να διαγραφεί. Μετά πάμε βέβαια και στον Φρόιντ που και ο Φρόιντ επίσημα μιλάει για έναν μηχανισμό απώλειας μνήμης και διερωτάται γιατί ξαφνικά αρχίζουν να χάνονται οι μνήμες των ανθρώπων. Ο Φρόιντ διερωτάται λοιπόν Ποιος είναι ο λόγος άραγε για τον οποίο οι ε, ασθενείς ξεχνάνε πάρα πολλά στοιχεία της ζωής τους και η απάντηση είναι η εξής. Όλα τα πράγματα που ξεχνάει κανείς ε, ίσως ήταν οδυνηρά ε, και κατόπιν τούτου ήταν φρικτά, επώδυνα και επονίδιστα. Το τραυματικό στοιχείο ανάγεται στο παρελθόν, οι επιπτώσεις όμως υπάρχουν και στο μέλλον στο παρόν με συγχωρείτε. Ε, πρόκειται για ένα παιχνίδι ανάμεσα στη μνήμη και την απώλεια μνήμης ε, και εναλλάσσονται αυτά τα δύο στοιχεία. Ένας άλλος πολύ σημαντικός ε, ήταν ο Γουλφεν Μπίον, ο οποίος μίλησε και αυτός για την απώλεια της μνήμης και μιλάει για ένα χρόνο ο, χωρίς ε, μνήμη, χωρίς επιθυμίες. Υπάρχει λοιπόν μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή πριν από τη μνήμη που έχει σχέση με το παρόν, με στιγμές του παρόντο, στιγμές όπου δεν έχει κανείς μνήμη του παρελθόντος και δεν έχει και εικόνες ε, για το μέλλον. Αυτό συμβαίνει όταν ε, παίζει κανείς ένα μουσικό όργανο ή όταν ε, τρέχει με τα θελτικά του παπούτσια ή όταν χορεύει με το ρυθμό του ταγκό. Τη στιγμή που βιώνουμε το παρόν βρισκόμαστε σε επαφή μόνο με συναισθήματα, με ασυνείδητη φάση ζωής αυτό λοιπόν το ασυνείδητο και τα όρια μεταξύ του συνειδητού και του ασυνείδητου, αυτά θα έπρεπε να είναι πάντα παρόντα ως διάφορα τμήματα της ε, νοητικής διεργασίας. Ε, είναι ε, ένα είδος κορεσμού της συνείδησης. Όμως θυμάμαι ε, και βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες ε, διαφάνειες ε, που προβάλλονται. Ας δούμε τι συμβαίνει όταν το παρόν καταστρέφει το παρελθόν και το μέλλον. Χάνονται τα συναισθηματικά βιώματα όπως η αγάπη, ο φόβος και έτσι λοιπόν φτάνουμε σε μια εναλλαγή καταστάσεων ε, χωρίς όμως να μπορεί κανείς να αφηγηθεί μια ιστορία, χωρίς να προκύπτει μια αυθόρμητη ιστορία. Είμαστε εκτός του γραμμικού χρόνου σε ένα συγκεκριμένο σημείο χωρίς συνέχεια. Είπαμε ότι δεν υπάρχει πλέον ιστορία, προκύπτει μια γενική αρχή. Ε, φτάνουμε κατά κάποιον τρόπο και στα όρια της αιωνιότητας. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά στην ασθένεια, υπάρχει και μια άλλη απώλεια μνήμης. Η οριστική απώλεια μνήμης, όπου ο άνθρωπος ε, μοιάζει να έχει χάσει την οντογέννησή του και η ε, ατομικότητά του γίνεται ασθένεια και προκύπτει ε, μια απήχηση που συγκαλύπτει τους, το πλαίσιο. Θυμούμαστε ξαφνικά πράγματα από το παρελθόν που είχαν όμως ε, ξεχαστεί τελείως και ξαφνικά ε, εκφράζονται διάφορα στοιχεία σαν άνθρωπος να μην είχε γεννηθεί ποτέ. Είναι λοιπόν ε, πολύ αδύναμο, αδύναμες αυτές οι διασυνδέσεις. Μιλάμε για τον εγκέφαλο ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργεί σωστά. Στην άνοια, εκείνος που υποφέρει ξεχ... έχει ξεχάσει ποιος είναι και χάνει τη συνέχεια της ζωής του. Πίνει το νερό της λύθης και βιώνει την άνοιά του. Προκύπτει ε, ένα χάσμα ανάμεσα στη συνείδηση του εξωτερικού κόσμου και του εσωτερικού. Η αρχική εικόνα ε, του εγκεφάλου είναι ένα παζλ, ένα μοσαϊκό από διάφορες εικόνες και το περιεχόμενο δεν ταυτίζεται με τις εικόνες. Είναι πραγματικά ένα ένιγμα αυτό. Ε, είναι σαν να υπάρχουν διάφορα μικρά καρτούν. Το μοσαϊκό αυτό ε, δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Πού τελειώνουν λοιπόν οι σκέψεις των ανθρώπων, οι ελπίδες τους, τα όνειρά τους, οι προσδοκίες τους, τα προγραμματά τους, οι επιλογές τους όταν γίνει η διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να συμβιώνουν με την ανασφάλεια, τη σύγχυση, τον αποπροσανατολισμό, την ανησυχία. Το άτομο δεν μπορεί να ε, ε, συνδεθεί με τίποτα, ούτε καν με το σώμα του. αποσυντίθεται, εφαλώς και ο άνθρωπος βρίσκεται σε, μια κατάσταση όπου υπάρχουν όλο και λιγότερες μνήμες. Ίσως κάποιες ε, μνήμες από τους οικείους, αλλά είναι ε, όλα αυτά ε, αποδιοργανωμένα. Χάνονται λοιπόν οι μνήμες στο κενό και διωγγώνεται όλο και περισσότερο αυτό το κενό. Οι συγκάτοικοι λοιπόν, οι συγκάτοικοι είναι εκείνοι που ζουν στον ίδιο οίκο της ασθένειας. Οι συγκάτοικοι μπορεί να είναι πολλοί, μπορεί να είναι και λιγότεροι, μπορεί να είναι ε, οι γιατροί, οι οικοί, αυτοί που τους ε, φροντίζουν. Αυτοί συγκατοικούν με την ε, άνοια και είναι αναγκασμένοι όλοι αυτοί να συγκατοικούν σε ένα χώρο όπου το άτομο παρετείται από την προηγούμενη αφήγησή του, από την δική του τη ζωή, από αυτό που συνέβη τη δική του με τη δική μας τη ζωή. Μιλάμε για τη δυστυχία των συγκατοίκων οι οποίοι ε, νιώθονται όλο και πιο δυστυχείς όταν δεν τους αναγνωρίζει ο Πάσχων. Ο πατέρας δεν αναγνωρίζει πλέον τα παιδιά του, οι, οι Εκείνη λοιπόν τη συγκεκριμένη στιγμή μετά τη διάγνωση τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει μία αμφισημία και δεν είναι εύκολο να ε, διαγνώσει κανείς ε, την αγάπη από άλλα συναισθήματα. Δεν αναγνωρίζει κανείς και το ε, σώμα του. Άρα δηλαδή προκύπτει μία αμφισημία όπως είπαμε και αυτή προκαλεί γενικότερα ανησυχία ανησυχία και στον ίδιο τον Πάσχοντα και στους ε, συγκατοίκους του. Ε, στην καθημερινότητα της ασθένειας δεν μπορώ να πω ε, πια τίποτα. Δεν μπορώ να πω ότι σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να πω δεν κατορθώνω ούτε καν να σε μισήσω. πρέπει να γυρίσω σε αυτό που ήμουνα παλαιότερα. Μπορώ να τα καταφέρω. Απάντησέ μου. Υπάρχει λοιπόν ε, αμφιβολία για όλα αυτά. Ο χρόνος γυρίζει στο ίδιο σημείο. Ε, ο ασθενής βρίσκεται πάντα μέσα στο κενό. Είναι αυτή, αυτές οι διακυμάνσεις των συναισθημάτων του ε, και με τον τρόπο αυτό προκύπτει μια αμφιθυμία. Ο ασθενής μπορεί να περνάει από ε, ανέκδοτα στον οργή ε, και όλα αυτά ε, είναι η έκφραση μιας ζωής που χάνεται. Ο συγκάτοικος πρέπει να αποσυνδεθεί από αυτό το, το κλειστό κύκλωμα. Και ποιες, ποιοι είναι οι κανόνες συγκατοίκησης τώρα για τους συγκατοίκους. Ε, στην σχέση με την ε, προοδευτική άνοια ε, προκύπτουν στιγμές όπου ο συγκάτοικος δεν γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Και για πρώτη φορά λοιπόν προσπαθεί να προκαλέσει βιώματα η δυσκολία των συγκατοίκων ή των οικείων να τους χαρακτηρίσουμε είναι σαφής, προσπαθούν να προκαλέσουν αισθήματα και αυτό προκαλεί ένα συγκάλυμα από το οποίο αναδύεται η αμφιθυμία ε, το άγνωστο για το άτομο, ε, το άγνωστο που καλείται ο Πάσχο να διασχίσει τα παιδιά ε, πρέπει να πενθήσουν για τον πατέρα ή για τη μητέρα που δεν υπάρχουν πια. Που ζουν βέβαια, αλλά δεν είναι άτομα. Έχουν θράψματα σε μιας εποχής που δεν επανέρχεται. Μέρα με τη μέρα λιώνει ο άνθρωπος και τελικά ε, ποιος θα ε, μπορέσει να κατανοήσει την κραυγή των παιδιών όταν δεν θα υπάρχουν πια οι γονείς. Δεν υπάρχει λοιπόν συνέχεια. Μιλάμε για την έλλειψη συνέχειας που ε, συνδέεται αυτή με την απώλεια της μνήμης. Και όταν θα πεθάνει ο Πάσχων θα είναι απλά ένας ακόμη θάνατος. Τα θράψματα της μνήμης θα οδηγήσουν στο ότι ε, δεν θα αισθάνεται κανείς ότι έχει μπροστά του τον άνθρωπο που γνωρίζει. Προσπάθησα να σας πω ε, πώς εγώ ε, μπορώ να υποσερμηνεύω την αμφιθυμία και την αμφισημία των ασθενών που νοσούν ε, από την ασθένεια Alzheimer. Και ίσως ε, να σας ε, δείξω ένα φιλμ, δεν είδα αυτό που προβλήθηκε προηγουμένως, είναι ένα φιλμ της Iris Murdoch, η συγγραφέας είναι Αγγλίδα, σεναριογράφος, ε, η ταινία είναι του 2001 και είχε Αλτσχάιμερ η σεναριογράφος ε, που διαγνώστηκε όμως μόλις το 2007 και το 2007 δημοσίευσε το τελευταίο της βιβλίο. Μια πολύ ζωντανή γυναίκα, ε, εγκεφαλική, για ανοιχτά και θέλησε να μιλήσει για την ελευθερία και για την αγάπη. Η ασθένεια την πλήττει και εκείνη που ζούσε πάντα αυτόνομη, αυτόνομα, δεν μπορεί πλέον ε, να ε, κινηθεί, χάνεται και ε, στο φιλμ τελικά ποιος ζει αυτό το δράμα της Άρης είναι ο Τζον ο σύζυγός της που μετά από 46 χρόνια γάμου με μια θαυμάσια γυναίκα έχει να κάνει μπροστά του με ένα ερωτηματικό Αισθάνεται λοιπόν ε, οργή, την απορρίπτει και αυτή είναι η αντίδραση. Γιατί δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε σχέσεις αγάπης. Η φυσιολογική αντίδραση είναι η οργή. Η οργή που μας ε, οδηγεί στο να απομακρυνθούμε από τους πάσχονες. Αυτό είναι το ε, συνηθισμένο. Όμως ε, ο Τζον αρχίζει να θυμάται και στην ταινία βλέπουμε το παρελθόν της Άιρης ε, που γίνεται και το παρόν διότι ο Τζον ε, έρχεται σε αντιπαράθεση με την Άιρης και γίνεται και αυτός ανοϊκός. Ε, ζούνε λοιπόν στο ίδιο σπίτι, τελικά το σπίτι είναι βρώμικο, κανείς δεν το καθαρίζει, τα βιβλία είναι άνω κάτω. Η ζωή λοιπόν των δύο ε, πρωταγωνιστών είναι αυτή. Τα βλία τα πετάνε παντού, στις σκάλες, παντού βρωμιά και μένουν ενωμένοι μέχρι το τέλος. Όμως ο Τζον σε αυτή την ε, φροντίδα ε, χωρίς σύνορα πενθεί. Πενθεί τη γυναίκα που υπήρξε και μετά το θάνατο της Άιρης θα γράψει δύο βιβλία για τη ζωή αυτής της γυναίκας. Υπάρχει και άλλη μια ταινία όπου ξεπερνιέται το ερωτηματικό. Είναι μια ταινία που προβάλλεται τώρα στη Βενετία. Είναι μια ταινία του Πούπια Βάτη ε, του Οκτωβρίου του 2010. Εκεί λοιπόν οι σχέσεις φροντίδας αντικαθίστανται γιατί δεν είναι πλέον μια ε, συζυγική αγάπη αλλά η πρωταγωνίστρια μετατρέπει τον σύζυγο που έχει άνοια σε μωρό που δεν μπόρεσε ποτέ να αποκτήσει. Και έτσι ζει μια πρωτογενή φροντίδα. Και ας δούμε λοιπόν τα συμπεράσματα. Γιατί είναι σημαντικό να μπορούμε και να καταθέσουμε μία πρόταση μετά από όλα αυτά που ελέγχθησαν. Τα συμπεράσματά μου λοιπόν είναι τα εξής. Ε, στις καθημερινές δυσκολίε ε, φροντίδας ε, ε, που σημαίνει ότι θα πρέπει κανείς να δείξει υπευθυνότητα και όλα τα συναφή ε, εναλλάσσοντας συναισθήματα, ε, οργή μεταξύ άλλων και ως εκ τούτου θα πρέπει κανείς να αναγνωρίσει τον πόνο που υπάρχει για την απώλεια, ένας, ένα πένθος και να αισθάνεται κανείς ότι χάνεται μία ζωή και εμείς δεν έχουμε την δυνατότητα να συσχετιστούμε με αυτή τη ζωή χωρίς ε, ερωτηματικά. Και θα ήθελα να αναφέρω την περίπτωση ενός ασθενούς ε, δικού μου που έκανε ανάλυση με μένα και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο ασθενής μου, χάνει τον πατέρα του από εγκεφαλικό και ο ασθενής μου δεν μπόρεσε να πενθήσει γιατί η μητέρα του ε, έχει Αλτσχάιμερ. Ο γιος λοιπόν δεν πάει ούτε στην κηδεία και τελικά ε, δεν κατορθώνει ούτε καν ε, να κλάψει και ε, περιτρέχει στην πόλη χωρίς να καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται. Προσπαθεί να κατανοήσει τι γίνεται και με τη μητέρα του που είναι κλινήρης. Κάποια μέρα λοιπόν η μητέρα, τον ασθενή μου το λένε Αντώνιο και η μαμά του δεν τον αναγνωρίζει. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή λέει στη μαμά του, ξέρεις ότι πέθανε ο μπαμπάς. Και λέγοντας το αυτό, ο Αντώνιο κατανοεί ότι πενθεί κατ' ουσίαν και γιατί τη μαμά που δεν υπάρχει πια, που τον ανέθρεψε, που τον γέννησε, που τον έκανε σημαντικό άνθρωπο. Και ο μπαμπάς έφυγε αλλά ο μπαμπάς δεν τον εγκατέλειψε, ο μπαμπάς πέθανε. Γι' αυτό λοιπόν εγώ επιμένω ότι το να επεξεργαστεί κανείς το πένθος, εδώ αναφέρομαι στους οικείους, αυτούς που χαρακτηρίζονται προηγουμένως συγκατοίκους, ε, το να ζήσουν αυτοί το πένθος είναι καθοριστική σημασία γιατί έτσι αποφορτίζεται κανείς, αποφορτίζεται και ζει μία κατάσταση η οποία παραλύει τους πάντες. Και πώς μπορεί να γίνει τώρα αυτό. Εγώ θεωρώ, επειδή είμαστε ε, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση 27 κρατών, όπως πες και ο κύριος Φριζόνη. Η δική μας η πρόταση είναι τα ε, νοσοκομεία, οι νευρολογικές κλινικές ε, να έχουν ένα ειδικό χώρο πτέρυγες, που να είναι πτέρυγες υποστήριξης και με ψυχαναλυτική υποστήριξη όπου ε, θα συντάσσονται κάθε φορά τα σχόλια να υπάρχει ένα είδος ε, ημερολογίου αν θέλετε σταματάει η να μιλάει ελέγχθη κάτι εκτός μικροφώνου κάτι αναφέρεται εκτός μικροφώνου Α, καλείται η ομιλήτρια να τελειώνει τέλειωσε Ευχαριστούμε κυρία Καπούτο. Thank you for your uh, interesting presentation from... Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ψυχοναλυτική προσέγγιση που μας παρουσιάσατε, αλλά σας πιέσα λίγο γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ε, ήταν λίγο μακροσκελέστερη η παρουσίαση σε σχέση με αυτά που περίμενα, οπότε θα ακούσουμε απευθείας τον καθηγητή Lars Όλοφο Βάλλοντ από το το τμήμα γυριατρικής ε, του Ινστιτούτου Καρολίνσκα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στο σημερινό εργαστήριο. θα ήθελα να συζητήσουμε κάποιες πτυχές της νόσου Αλτχάιμερ και της άνιας. Ένα συνδυασμός του τι συμβαίνει στον ασθενή, και ε, το πώς επηρεάζει αυτό τους οικείους του. Και επίσης θα σας μιλήσω λίγο και για την πρόληψη. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Λοιπόν, ε, θα σας μιλήσω για τα συμπτώματα της συμπεριφοράς και τα ψυχιατρικά συμπτώματα που είναι γνωστά με το αγγλικό ακρονίμιο BPSD. Είναι μη γνωσιακά συμπτώματα, δεν αφορούν στη μνήμη και επέρχονται κατά περιόδους ε, κατά την εξέλιξη της νόσου και δημιουργούν μεγάλο άγχος και στον ασθενή και στους περιθάλποντες ε, και οφείλονται κατά πάσα πιθανότητα στη ζημιά που έχει υποστεί ο εγκέφαλος ε, και οι διαβιβαστές. Αλλά δεν είναι αυτά καθεαυτά η αιτία ε, η εξήγηση μπορεί να αναζητηθεί στην ε, διάδραση ανάμεσα στο περιβάλλον, τον ασθενή και τους περιθάλποντες. Πώς ερμηνεύει δηλαδή το περιβάλλον του ο ασθενής. Ε, η ερμηνεία που δίνει οδηγεί και στην εμφάνιση των συμπτωμάτων. Συγκεκριμένα παραδείγματα αυτών των συμπτωμάτων είναι η κατάθλιψη, στα αρχικά στάδια της εξέλιξης, παρεστήσεις, παραλυρήματα, επιθετική συμπεριφορά, άσκοπη υπερυπλάνηση, υπερπατούν 8-10 ε, ώρες μέσα στη μέρα οι ασθενείς, ε, ε, δημιουργεί αυτό μεγάλο άγχος, διαταραχές του ύπνου, αγωνία, απάθεια. Και ορισμένα είναι που δημιουργούν μεγάλο άγχος και άλλα συμπτώματα λιγότερο άγχος, Βλέπετε εδώ το σχήμα εξέλιξης ε, της νόσου ε, για μια περίοδο 10-15 ετών. Στα αρχικά στάδια, στα αριστερά δηλαδή του διαγράμματος, βλέπετε την ε, κατάθλιψη, το άγχος στο, στα μεσαία στάδια της παρεστής και τα παραλυρήματα και κατόπιν με υψηλό άγχος φυσικά η επιθετική συμπεριφορά και η άσκοπη περιπλάνηση. Ε, πώς μπορεί κανείς να θεραπεύσει αυτά τα συμπτώματα. Όταν άρχισα την ε, καριέρα μου στο τμήμα γυριατρικής υπήρχε μία μόνο θεραπευτική αγωγή ή φαρμακολογική αγωγή. Φαρμακευτική συγγνώμη αγωγή. Ε, τώρα προσπαθούμε να μην αρχίζουμε με αυτή την αγωγή, αναζητούμε τα αίτια των συμπτωμάτων. Ανά, υπάρχει κάτι ανάμεσα στον ασθενή και στους περιθάλποντες ή στη σχέση του με το περιβάλλον. Ε, άλλες ε, θεραπείες ε, είναι η θεραπεία της αποδοχής, η ανάκληση των αναμνήσεων και άλλες θεραπευτικές αγωγές. Όταν τα έχουμε δοκιμάσει όλα αυτά χωρίς επιτυχία, τότε μπορούμε να περάσουμε στη φαρμακευτική αγωγή. Έχουμε νέες κατευθυντήριες γραμμές στη Σουηδία για τη θεραπεία και τις κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Ινστιτούτου για τους ασθενείς που πάσχουν από άνοια. Ε, και βλέπουμε ότι δεν είναι η πρώτη επιλογή η φαρμακευτική αγωγή. Τώρα, φαρμακολογική αγωγή. Ε, χορηγούμε χαλοπεριντόλ παραδείγματος χάρη ε, και άλλα φάρμακα κατά της άνοιας, ε, τους ε, αναστολίσα και τυλχολινεστεράζεις, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν και εναλλακτικέ θεραπείες, αλλά δεν έχουμε ισχυρά τεκμήρια για τα αποτελέσματά τους. Η ανάκληση των αναμνήσεων χρησιμοποιείται κατά κόρον αλλά χρειάζεται πολύ ευρύτερη έρευνα για να αποφασίσουμε τι συνιστά καλή θεραπευτική αγωγή. Επόμενη διαφάνεια η συστηματική αναθεώρηση των θεραπείων ε, δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Ποιος ήταν ο στόχος ε, να έχουμε πολλές δημοσιεύσεις για τις μη θεραπευτικές αγωγές. 179 ε, το αριθμό τελικά. 179 δημοσιεύσεις, χαμηλότερες ή υψηλότερες ποιότητες. Ε, οι παρεμβάσεις που χρησιμοποίησαμε για την κατάταξη σε ήταν γνωσιακή εκπαίδευση, διάφορα γνωσιακά ρεθίσματα, ανάκληση αμνήσεων, η χρήση φωτός, αποδοχή και για τους περιθάλποντες η εκπαίδευση, η υποστήριξη, η φροντίδα εκτός οικίας κτλ. Ε, ε, κάποια αποτελέσματα κατεδείχθη ότι οι περιθάλποντες, μάλλον ε, έχουμε μια πολύ ε, παραγωγική παρέμβαση για τους περιθάλποντες. Ε, ανάλογα μιλάμε για κέντρα περίθαλψης, το 1 τρίτο των ασθενών, αν γίνεται περίθαλψη κατοίκων. και τώρα, θετικά αποτελέσματα έχουμε με την γνωσιακή εκπαίδευση, την εκπαίδευση ADL, την πολυπαραγοντική παρέμβαση και αμφισβητούμενα είναι τα αποτελέσματα της ανάκλησης των αναμνήσεων, της ψυχαγωγίας κτλ. Κατόπιν, υπήρχε ένας υψηλός αριθμός παρεμβάσεων που δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Γιατί, διότι δεν υπήρχαν αρκετές ε, μελέτες, ε, ε, μέτρα για να εφαρμοστούν τα αποτελέσματα αυτών των μελετών και αυτά φαίνονται στην ενδιάμεση αναθεώρηση που δημοσιεύθηκε. Για να περάσουμε στο άγχος των περιθαλπώντων, είναι μια άλλη πτυχή της άνοιας. Οι οικοί περιθάλποντες Ακούσαμε ήδη σήμερα ότι πλήττονται σοβαρά από την ε, άνοια. Γνωρίζουμε ότι οι περιθάλποντες ε, των ασθενών ε, παρουσιάζουν σημάδια κατάθλιψης, άγχους, αϊπνίας, και άλλες ψυχοσωματικές παθήσεις. Εδώ πέρα έχουμε περισσότερα επιστημονικά στοιχεία, η ψυχοεκπαίδευση, υποστήριξη από ομάδες συμπασχόντων, η ψυχολογική θεραπεία, κυρίως όταν είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες ε, της συγκεκριμένης περίπτωσης, οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα και μπορεί να μειώσει το άγχος των περιθαλπόντων. Επίσης, ε, από τα, την Ένωση των κέντρων, ε, ημερησίων κέντρων περίθαλψης έχουμε κάποια στοιχεία, εν συντομία να σας πω, και το ακούσαμε και νωρίτερα, ότι οι περιθάλποντες ε, καταναλώνουν πολύ χρόνο για την περίθαλψη των συγγενών τους, κυρίως όταν πρόκειται για ασθενείς άνοιας, πάνω από 4-5 ώρες την εβδομάδα αφιερώνονται στην περίθαλψη την εβδομάδα. Επόμενη διαφάνεια σας είπα ποια είναι τα αποτελέσματα στην υγεία. Έχουν αυξημένη πίεση, επίπεδα ενσουλίνης, ε, ανεπαρκή νοσοποιητικά συστήματα, αυξημένο κίνδυνο για καρδιακιακές ε, παθήσεις. Ε, επίσης, υψηλή θνησιμότητα, κατά 63%. Ε, γνωρίζουμε ότι οι περιθάλποντες των ανοικών κατά 40% ε, ε, υποφέρουν από κατάθλιψη και από άγχος. Ένα παράδειγμα για μια μελέτη παρέμβασης 229 ε, περιθάλποντες ε, μελετήθηκαν ε, με ενισχυμένη υποστήριξη και συμβουλές για έξι συναντήσεις. Αυτή η μειωμένη, μειωμένη κλίμακας παρέμβαση οδήγησε σε λαντωμένα συμπτώματα κατάθλιψης. Έχουν, έχει πολύ ευεργετικό αποτέλεσμα με τέτοιου είδους παρέμβαση δηλαδή στους περιθάλποντες. Τέλος, πρόληψη. Όπως είπε η κυρία Φρυσόνη, ε, έχουμε αποτελεσματικές φαρμακευτικές αγωγές και συνεχίζουμε να ζητούμε την βέλτιστη δυνατή αγωγή ε, αλλά χρειαζόμαστε και αυξημένε γνώσει για την πρόληψη τη νόσου. Γνωρίζουμε από επιδημιολογικέ ε, μελέτε ότι η υψηλή ε, κατανάλωση ψαριών μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο κίνδυνο για εμφάνιση τη νόσου Αλτσχάιμερ. Ε, μία μελέτη που κάναμε στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα πριν από κάποια χρόνια ε, και ονομάστηκε η μελέτη ωμεγα 3, λιπαρών οξέων δηλαδή, για, 6, για 9 μήνες ε, κατέδειξε ότι αυτοί που είχαν ότι υπήρχαν θετικέ επιπτώσεις από την υψηλή κατανάλωση ψαριών και είχαν βελτιωμένες ε, λειτουργίες ε, μνήμης, παραδείγματος χάρη, ή μνήμη, παραδείγματο χάρη, μικρότερη γνοσία ε, επίσης άλλη μελέτη η οποία ονομάζεται Lipd Diet τώρα άρχισε και εξετάζεται η γνωσιακή ανεπάρκεια στα αρχικά της στάδια σε 300 ασθενείς με χρήση εικονικών φαρμάκων ή με ένα κοκτέιλ φαρμάκων που συμπεριλαμβάνει και τα λιπαρά οξέα ωμέγα 3. Αυτές οι δύο μελέτες λοιπόν, να περάσουμε στα συμπεράσματα. Ξέρουμε ότι αυτά τα συμπτώματα, τα BPSD, ε, είναι πολύ κοινά, σχεδόν όλοι οι πάσχοντες ε, τα εμφανίζουν, δημιουργούν μεγάλο άγχος και για τους ασθενείς ε, και για τους περιθάλποντες. Τώρα, κατά προτεραιότητα προτιμούμε τις μη φαρμακευτικές αγωγές, αλλά θέλω να το τονίσω, για να βρούμε τι αποτελεσματικότερες θεραπευτικές αγωγές χρειάζεται εκτεταμένη έρευνα. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι περιθάλποντες ε, έχουν υψηλό κίνδυνο για ε, ψυχοσωματική νοσηρότητα και άρα χρειάζεται ε, εκτεταμένη έρευνα για να βρούμε τις κατάλληλες μεθόδους και για να έχουμε και τα απαιτούμενα μέσα ώστε να είναι αποτελεσματικές οι παρεμβάσεις που κάνουμε και επίσης χρειάζεται έρευνα για το, την τροφή που χρησιμοποιείται ως φάρμακο ε, για την ε, εκρίζωση της νόσου σε κάποιες ομάδες ασθενών ε, και για την πρόληψη της κυρίως. Ε, αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με το πάνελ, με όλους τους προσκεκλημένους μας δηλαδή. Τώρα πριν ζητήσετε το λόγο, να σας πω ότι αν έχουμε χρόνο αργότερα θα επανέλθουμε στην παρουσίαση της έκθεσης της κυρίας Μάτιας και θα πάρουν το λόγο οι σκιώδες. Λοιπόν, τώρα ερωτήσεις, αλλά όχι επί της έκθεσης, αυτό θα γίνει αργότερα. Ε, κάντε ερωτήσεις μόνο στους προσκεκλημένους. Η κυρία Αντωνέσκου έχει το λόγο. Ξέρω ότι είσαστε σκιώδης από το για την έκθεση μάτιας, αλλά επαναλαμβάνω ερωτήσεις στο πάνελ μας και προσδιορίστε σε ποιον απευθύνεται την ερώτησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να αναφερθώ στον κοινό προγραμματισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων. Δυστυχώς δεν ήμουν εδώ από την αρχή σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω για την οργάνωση του εργαστηρίου μας και ευχαριστώ πολύ όλους τους προσκεκλημένους για τις παρουσιάσεις τους. Έτσι, δεν μπορούσα να ακούσω την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ θέλω να αναφερθώ στο κοινό προγραμματισμό ερευνητικών δραστηριοτήτων. Και αυτό γιατί για μένα είναι το πιο σημαντικό βήμα που μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να καταπολεμήσουμε αυτή την ασθένεια. Ποιο είναι το ποσοστό χρηματοδότησης λοιπόν διακόπτη η Πρόεδρος. Το ερωτηματικό δεν βλέπω. Βάλτε ερωτηματικό παρακαλώ. Ερώτηση να κάνετε και σε δύο λεπτά μόνο, όχι παραπάνω. Μετά θα ξανέχετε το λόγο Σκιώδης. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Αντωνίσκου. Ρωτάω λοιπόν, ποια είναι η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σχέδιο αυτό για συμπρογραμματισμό, από κοινού προγραμματισμό. Πόσο συμμετέχει στη χρηματοδότηση, αυτό θέλω να ξέρω. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, θα σας απαντήσω. Γιατί είδατε ο κύριος Φαί έπρεπε να φύγει. Το στην αρχή. Ήταν ο πρώτος ομιλητής, ήταν πολύ ξεκάθαρος. Και θα φροντίσει η Επιτροπή να απαντηθεί το ερώτημα της κυρίας Αντωνέσκου. Και στον επόμενο γύρο συζητήσεων θα επανέλθουμε σε αυτό. Επόμενος, ο κύριος Γιωβάνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ρωτήσω. Μήπως νομίζετε κι εσείς ότι η ευρωπαϊκή έρευνα χρειάζεται λιγότερο κατακαιρματισμό και ότι οι διάφοροι ειδικοί που ενδιαφέρονται για το Αλσχάιμερ να μπορούν από κοινού να δουλεύουν. Δεν θα ήταν πιο αποτελεσματικό. Είτε πρόκειται για τους κεταρολόγους είτε πρόκειται για βιοχημικούς, είτε πρόκειται για ψυχολόγους, για κλινικούς γιατρούς όλες αυτές οι ειδικότητε. Δεν θα έπρεπε μαζί να συνεργαστούν. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ναι, μεν τα μέσα υπάρχουν, αλλά είναι κατακαιρματισμένα και γεωγραφικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, μεταξύ διαφόρων ειδικοτήτων. Δεύτερον, μιλήσατε κι εσείς για την αμαλουδή πρωτεΐνη. Η ερώτησή μου είναι απλή. Έτσι όπως ξέρουμε τα πράγματα σήμερα, δεν έχετε την αίσθηση ότι η πρωτεΐνη αυτή αποτελεί σύμπτωμα της ασθένειας και όχι την αιτία της. Μπερδεύομαι λίγο με την παρουσίασή σας. Διότι από αυτά που έχω διαβάσει φαίνεται ότι μπορούμε με να περιορίσουμε τα αμυλοειδή, αλλά δεν έχουμε κλινική αλλαγή. Οπότε αυτό δεν θυμίζει λιγάκι την περίπτωση καρκίνων που προκαλούν εμετούς, διορθώνουμε τους εμετούς, τους αποφεύγουμε, αλλά δεν θεραπεύουμε τον καρκίνο. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Πριν απαντήσετε, μια που έχουμε άλλη μια ερώτηση από τους ευρωβουλευτές, σας την ακούσουμε και αυτήν, τη Λίντα Ματκάβεν, και μετά να απαντήσετε. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον τελευταίο μιλητή όσον αφορά την πρόληψη. Αναφερθήκατε στο Μέγα 3, την τροφή. Πόσο αλήθεια είναι. Αν όντως έχει ουσία αυτό που λέτε, είναι πράγματι έτσι, είναι κάτι που το ξέρει ο κόσμος, που είναι ευραίος γνωστό πια, ή είναι περιορισμένο έτσι σε κάποιο ερευνητικό, πρόγραμμα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, αν όντως είναι αλήθεια, στέκει και είναι ευραίος γνωστό, πρέπει να αλλάξει ο κόσμος συνήθειες διατροφής. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Λέει η κυρία τρει τρεις ερωτήσεις. Συμφωνώ και με αυτά που είπε ο κύριο Ζουβά, με τη δικιά του ερώτηση. Δηλαδή, η ευρωπαϊκή έρευνα πρέπει να, έχει, να δίνει κάτι παραπάνω. Οι ερωτήσεις μου είναι προς τον δόκτωρα Φρυσόνη. Πιστεύετε ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι έρευνε σήμερα είναι ικανοποιητικό ή θα έπρεπε να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες. Θέλουμε να βρούμε ένα φάρμακο που είτε να θεραπεύει είτε να βελτιώνει την κατάσταση των ασθενών. Αλλά για να το κάνουμε αυτό δεν θα έπρεπε το εύρος των ερευνών να είναι μεγαλύτερο. Εγώ δεν είμαι γιατρός, οπότε δεν ξέρω πολύ από αυτά. Δεν θέλω να μπω στα ιατρικά επιχειρήματα, αλλά από αυτά που διαβάζουμε είναι μήπως δεν πρέπει να περιοριστούμε στην αμυλοειδή πλάκα, αλλά να διευρύνουμε περισσότερο τις έρευνές μας. Κάτι άλλο τώρα για το ωμέγα 3. Και μένα με απασχολεί πολύ αυτό, αλλά με απασχολεί και το θέμα του καπνού. Υπάρχει μια μελέτη στη Φιλανδία που μόλις δημοσιεύτηκε, που πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Εκεί διαβάζουμε ότι φαίνεται ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στους μεγάλους καπνιστές, δηλαδή πάνω από τρία πακέτα την ημέρα, ότι αυτοί έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να πληγούν από Αλσχάιμερ. Εσείς τι γνώμη έχετε για αυτού του είδους τις έρευνες. Ευχαριστούμε. Για να ρίξω μια ματιά, λέει πρόεδρο, μήπω είναι κανένα άλλο. Όχι, δεν βλέπω άλλη ερώτηση. Οπότε θα δώσω το λόγο στου δύο, στου οποίου απευθύνθηκαν ερώτηση. Δεν ξέρω, Φασόνη, Βόλιν, ποιο από του δύο. Κύριε Φασόνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις ερωτήσεις κυρία Πρόεδρε. Μπορώ έτσι να εξηγήσω αυτά που δεν μπόρεσα να εξηγήσω λόγω του περιορισμένου χρόνου που είχα. Ο κατακαιρματισμός της έρευνας στην Ευρώπη. Εννοείται, εννοείται. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι δεν πρέπει να υπάρχει κατακαιρματισμός. Γι' αυτό και υπάρχει η πρωτοβουλία για τον κοινό προγραμματισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ, ότι για να έχουμε ένα αρμονισμένη επιστημονική έρευνα στην Ευρώπη πρέπει να έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Οι επιστήμονες πρέπει να έχουν μια ονομασία. Ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα. Στις Ηνωμένε Πολιτείε και συγγνώμη που πάντα θυμίζουμε τι γίνεται από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, αλλά τι να κάνουμε. Δουλεύουμε σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Άρα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τι γίνεται κι αλλού. Στις Ηνωμένε Πολιτείε λοιπόν μπόρεσαν να αναπτύξουν ένα τεράστιο, φιλόδοξο πρόγραμμα και ξεκινάνε με το φιλόδοξο αυτό για το επόμενο στάδιο. Πρώτα ήταν για τη μνήμη, τώρα περνάνε στο επόμενο στάδιο. Πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος εννοείται. Και αυτό για να απαντήσω και στην ερώτηση της κυρίας. Λυπάμαι, αλλά το όνομά της μου διαφεύγει. Πρέπει να βρείτε, να εντοπίσετε τον κατάλληλο χώρο έρευνας. Συμφωνώ. Τώρα είμαστε στις δομές για τους ερευνητές. Εκεί υπάρχει ο χώρος. Στο γενικότερο σενάριο, ορισμένες χώρες δεν δίνουν κονδύλια γι' αυτό. Εκείνη λοιπόν που πρέπει να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. για τον ρόλο των αμυλοειδών. Δεν μπήκα σε λεπτομέρειες. Εγώ ανέφερα και τα πεπτίδια και τα αμυλοειδή. Δεν θα μπω τώρα, εγώ δεν είμαι βιολόγος. Όμως υπάρχει ευρία συνένεση μεταξύ των επιστημόνων ότι πρώτα έρχονται τα αμυλοειδή και μετά η νευροεκφυλιστική συνέχεια. Τώρα, τι είναι ανάμεσα στα δύο. Τα αμυλοειδή συγκεντρώνονται σε κάποιους χώρους των εγκεφάλων και τα νευροεκφυλιστικά φαινόμενα τα βρίσκουμε σε κάποια άλλα σημεία του εγκεφάλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα αμυλοειδή αποτελούν μόνο σύμπτωμα της ασθένειας. Οι οικογένειες, αυτό Τώρα καταλήγουμε σε επιστημονική συζήτηση εδώ και δεν θα θέλαμε. Αλλά τέλος πάντων. Καλά, θα σταματήσω, θα σταματήσω. Εντάξει. Α, ευχαριστώ πολύ κύριε Φασόνη. Ο κύριος Ζουβά. Διμερός θα μπορούσε να κάνει αυτή την ιατρική συζήτηση με τον κύριο Φρυσόνη. Τώρα, ο καθηγητής Βαλάν. Ξέρω ότι και άλλοι όμως από το πάνελ θέλουν να απαντήσουν Μετά θα κάνουμε και τα λίγα πόσο για την έκθεση, οπότε πρέπει να προχωράμε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, με ρωτήσατε για το ω3. Από τα δεδομένα που έχουμε, που είναι νέα, είναι επιδημιολογικές μελέτες που πρέπει να ξέρουμε ότι κρατάνε 10-12 χρόνια προκειμένου να ξέρουμε αν κάτι Όντω είναι έτσι όχι. Οι πρώτες κλινικές μελέτες μόλις έχουν ξεκινήσει. Και αυτό γιατί οι δοκιμές κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα. Είναι πολύ λίγες οι επιχειρήσεις, οι εταιρείε που χρηματοδοτούν αυτές τις μελέτες. Άρα, τις κλινικές μελέτες. Άρα είμαστε στην αρχή μόνο με τις βιταμίνες. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώ. με αυτές τις ουσίες πρέπει κανείς να ξεκινάει πολύ νωρίς. Στα αρχικά στάδια. Για το κάπνισμα τώρα επίση με ρωτήσατε. Αν είναι βλαβερό. Ναι, είναι. Οι μελέτες δείχνουν ότι το πολύ κάπνισμα αυξάνει τις πιθανότητες να αναπτύξετε ασθένειες, άνοια ή αλσχάιμερ. Προχωράμε και εντοπίζουμε όλο και περισσότερο ομάδες κινδύνου και οι καπνιστές που καπνίζουν πολύ, όντως, φαίνεται να περιλαμβάνονται εκεί. Είναι πολύ σημαντικό πράγματι να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε ομάδες κινδύνου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Παρακαλώ. για το συντονισμό των ερευνητικών προσπαθειών, λέει εκπρόσωπος της Alzheimer. Χρειάζονται όντως και περισσότερες μελέτες, αλλά και καλύτερα συντονισμένες. Εμείς χαιρόμαστε πολύ λοιπόν που υπάρχει αυτή η κοινή πρωτοβουλία, η πρωτοβουλία για το κοινό πρόγραμμα δηλαδή. Έτσι ώστε να ξέρουμε και τι έρευνες χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο. Εδώ και 6 μήνες έχουμε ξεκινήσει, αλλά ακόμα δεν έχουμε την απάντηση απόλυτα. Οπότε, χρειάζεται πράγματι καλύτερο συντονισμός για να ξέρουμε τι ερευνητικέ δραστηριότητε λαμβάνουν χώρα. Και το τελευταίο που έχω να πω είναι το εξή. Δεν πρέπει να είναι μόνο η ιατρική έρευνα αυτή. Ελπίζουμε εμείς οι οργανώσεις ασθενών Αλτσχάιμερ ότι κάποια στιγμή θα έχουμε την πρόληψη, τη θεραπεία. Αλλά πρέπει σήμερα έτσι όπως έχουν τα πράγματα να μπορούμε και να ανταλλάσσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, να ανακουφίζουμε τους ανθρώπους και να υπάρχει τρόπος χρηματοδότησης για αυτούς που φροντίζουν τους πάσχοντες. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Ευχαριστούμε. Η κυρία Λί. Παρακαλώ γρήγορα κυρία Ευχαριστώ. Είμαι πρόεδρος της ε, αντίστοιχης οργάνωσης εδώ στο Βέλγιο. Πρέπει να σας πω ότι εκπροσωπώ τις οικογένειες, τους πάσχοντες και έχουμε βρει βοήθεια, όχι βέβαια αρκετή, από τα διάφορα δίκτυα. Τα δίκτυα που δουλεύουν στην έρευνα και την ψυχολογική και την κοινωνική είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η ανταλλαγή απόψεων μαζί τους είναι προτεραιότητά μας. Όμως αυτό που επίσης πιστεύω πολύ σημαντικό και θέλω εδώ να το υπογραμμίσω δεν είναι ότι επειδή κάποιος πάσχει από Αλσχάιμερ δεν εξακολουθεί να είναι άνθρωπος μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής του και παραμένει ένας άνθρωπος που αγαπάμε και αγαπάει ακόμα και αν εκφράζεται διαφορετικά. Και επιμένω πάνω σε αυτό γιατί το έχω ζήσει και εγώ. Γίνεται. Και το λέω για όλους αυτούς που ασχολούνται με τους πάσχοντες ότι πρέπει να έχουν κουράγιο και δύναμη να δούνε τον άνθρωπο αυτό σαν έναν άνθρωπο τον οποίο φροντίζουμε. Και δεν πρόκειται για ένα αντικείμενο που φροντίζουμε, αλλά για έναν άνθρωπο μέχρι το τέλος της ζωής του. Ήρθε εκπρόσωπος Επιτροπής ο κ. Φαΐ, οπότε σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε στην ερώτηση της κυρίας Αντωνέσκου. Λεπτομέρειες γραπτά, αν θέλετε, εφόσον σκοπεύετε να μιλήσετε πάνω από δύο λεπτά, αλλά αν σε δύο λεπτά μπορείτε να απαντήσετε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ξέρετε ότι στην Επιτροπή ασχολούμαστε με πολλά και διάφορα θέματα. Επειδή στην υγεία δεν είμαστε πολλοί, γι' αυτό και διαχειόμαστε πάμε από ένα μέρο στο άλλο. Γι' αυτό και έλειψα. Πάντως, για την ερώτησή σας, για το εύρος της έρευνας. Έχουμε την τάση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικεντρώμαστε σε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το πιο χρήσιμο, που είναι θεμελιώδης έρευνα. Όμως ένα από τα πράγματα που ακούω πρόσφατα είναι ότι πρέπει να έχουμε μια συνολική προσέγγιση, ολιστική, για να μπορούμε τα επιμέρους αποτελέσματα ερευνών να τα συμπεριλάβουμε σε ένα γενικότερο σύνολο. Εδώ βέβαια είναι και το Συμβούλιο που μπαίνει μέσα. Είπαμε πριν ότι δεν φτάνει να δούμε ένα συγκεκριμένο άτομο πώς αντιμετωπίζεται, τι του χρειάζεται. Για την πρωτοβουλία και την ε, καινοτομία όσον αφορά την γύρανση του πληθυσμού, Θέλω να τονίσω ότι είναι προς το συμφέρον όλων όσοι συμμετέχουν εδώ σήμερα να παρακολουθήσουν από κοντά αυτή την πρωτοβουλία. Συνεχίζουμε να την ολοκληρώνουμε, έτσι η διαβούλευση συνεχίζεται. Και ο πρόεδρος Μπαρόσο και όλοι οι επίτροποι ενδιαφέρονται πολύ για αυτή την πρωτοβουλία. Ελπίζουμε ότι θα στηριχτεί και οικονομικά. Γιατί θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την καινοτομία Ακριβώς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα ζητήματα που τέθηκαν στη συζήτηση εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε. Το πήραμε το μήνυμα ότι χρειάζεται πίεση από εμά και στήριξη. Το καταλάβαμε. Σίγουρα η συγκήτρια με τους σκιώδες εισηγητές θα φροντίσει στην έκθεση να συμπεριληφθεί αυτό και ενδεχομένω να υποβάλουμε τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ωραία, τελειώσαμε και με το δεύτερο τμήμα του εργαστηρίου μας. Ερχόμαστε στο τρίτο τμήμα που είναι ευρωβουλευτές που συζητούν για την ε, Άνια. Εδώ θέλω να σας πω και τη δικιά μου την εμπειρία λιγάκι. με εδώ 21 χρόνια. Πάντα σχολιόμουν με την υγεία, με τα τρόφιμα, με τις παρελβοντικές ε, πολιτικές η υγεία ήταν πάντα πολύ πιο κοντά σε μένα και προσπαθώ τώρα εδώ να μην συγκινηθώ με αυτά που λέω. Ασχολήθηκα με τις ασθένειες εκείνες που πολλές φορές δεν είναι τόσο γνωστές στο ευρύ κοινό. Μια τέτοια κατηγορία ήταν οι ασθένειε όπω η Άνια, οι ψυχικές ασθένειες. Πριν από 8 χρόνια πέθανε ο πατέρας μου από καρκίνο σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Η μητέρα μου ζει μόνη τη. Μάλλον ε, ζούσε μόνη τη, Την έχασα τον Ιανουάριο. Ήταν 79 ετών, ήταν σε καλή φυσική κατάσταση. Κάποια στιγμή άρχισε να μου φαίνεται περίεργη και δεν καταλάβαινα τι ακριβώς ήταν το περίεργο πάνω της. Άρχισε να συμπεριφέρεται περίεργα. Παλιά ήταν κι άλλη μέσα στο σπίτι. Τώρα που έμενε μόνη της, ξαφνικά άρχισε να χάνει πράγματα. Και της έλεγα, Μα δεν είναι δυνατόν, αφού μόνη σου ζεις εκεί, πώς τα έχασες. Κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Πέρασε πολύ καιρό μέχρι να καταλάβω ότι είχε κάποια μορφή άνοιας. Ενάμισης χρόνος χρειάστηκε. Πέρασαν δέκα μήνες Ενάμεσα στα συμπτώματα και την διάγνωση. Ζαν, άκουσα την παρουσίασή σου τι είπες για τη Γερμανία. Ε, ειδικά με εμπειρία διαφορετική στη Γερμανία. Χρειάστηκα περισσότερο χρόνο. Ήθελε πάντα να το κρύβει όμως η μητέρα μου ότι είχε άνοια. Έλεγε ότι υπάρχει μια τρικυμία στο μυαλό μου. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό βέβαια. Θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι δεν είχε κάποιον όγκο, γιατί αυτό σκεφτήκαμε στην αρχή. Κάναμε ένα σκάνινγκ και τη είπαν, όχι, όχι, δεν έχετε κανέναν όγκο. Και ήταν ενθουσιασμένη, είπα, δεν έχω τίποτα, είμαι μια χαρά. Ο νευρολόγος, γιατί δεν ήθελε η μητέρα μου να πάω σε κάποιον ειδικό, μου είπε ότι είχε κάποια ατροφία ενός τμήματος του εγκεφάλου. Ε, υπήρχε ένα τμήμα που μεγάλωνε και που πίεζε άλλα τμήματα του εγκεφάλου. Πήρε φάρμακα γιατί ήθελε να πάρει φάρμακα, αλλά μου είπε ο νευρολόγος ας τα πάρει τα φάρμακα, αλλά ό,τι και να κάνει να ξέρει ότι δεν θα έχει διαφορά η εξέλιξη. Συνέχισε να μόνη της. Αλλά αλλάξαμε την κλειδαριά, την πόρτα της εισόδου, τέσσερις φορές μέσα σε λίγους μήνες, γιατί τέσσερις φορές έχασε τα κλειδιά της. Ήταν 78 Έμοιαζε όμω σαν να ήταν 65, γιατί ήταν αδύνατη, έτσι έδειχνε δυνατή, σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Εγώ το έβλεπα ότι κάτι πολύ άσχημο συνέβαινε όταν το 2009 ξέχασε τα γενέθλιά μου. Εγώ δεν την πήρα τηλέφωνο να της πω «Μαμά, είναι τα γενέθλιά μου, γιατί δεν με πήρες να μου πεις χρόνια πολλά». Αλλά κατάλαβα ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Όλο όσα είπε η δόκτωρ Καπούτο δεν τα κατάλαβα με τη μητέρα μου. Είναι πολύ ψυχοαναλυτικά αυτά που μας είπε. Αλλά το να χάνεις κάποιον ή να αναγνωρίζεις ότι κάποιος είναι μεν ζωντανός αλλά τον χάνεις από αυτό που ήταν πριν, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους. Μπορεί να είσαι πολύ μορφωμένος, μπορείς να γνωρίζεις ένα σωρό πράγματα για το θέμα, παρόλα αυτά πονάει πολύ. Έχω την εντύπωση για τον εαυτό μου ότι είμαι καλά ενημερωμένη, μορφωμένη, παρόλα αυτά δεν ήξερα πώς να αντιμετωπίσω Πήρα το ζωσά και το Εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα. Πάντως, ώστε να έχουμε πολύ γρήγορα διάγνωση μετά από τα πρώτα συμπτώματα. Και να ξέρουμε ποια είναι αυτά τα πρώτα συμπτώματα είναι πολύ σημαντικό. Η Άννα και εγώ, τώρα που ακούγαμε τις παρουσιάσεις, κοιταζόμαστε και λέγαμε «Όχ, και εγώ ξεχνάω ονόματα, όχ, και εγώ έχω χάσει το κινητό μου, πρέπει να ανησυχώ». Είναι άνοια. Σε όλους συμβαίνουν ε, τέτοια πράγματα. Αλλά αν είναι επαναλαμβανόμενα, μπορείς να πας σε ένα γιατρό. Αμέσως αμέσως ξέρεις ότι δεν είναι κάποια άλλη αρρώστια, για παράδειγμα, ότι δεν είναι καρκίνος, ότι δεν είναι κάτι. Συνήθως όταν ε, έχουμε την καρδιά μας, πίεση και αυτά, πάμε στο γιατρό με τα πρώτα συμπτώματα. Με τα πρώτα συμπτώματα της άνοιας όμως δεν πάμε, γιατί δεν τα αναγνωρίζουμε. Η κυρία Ντονέσκου μίλησε για την έρευνα. Ναι, όντως η έρευνα είναι το πιο σημαντικό, αλλά το άλλο σημαντικό είναι η Alzheimer Europe και όλες οι οργανώσεις και ενώσεις για το Alzheimer τι κάνουν, να ενημερώνουν τον κόσμο, να του εξηγούν ότι υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης. Τώρα που έχουμε ψηφίσει τη διασυνοριακή υγεία στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια ελπίζω θα περάσει, μπορεί κανείς να πάει αλλού για θεραπεία. Στη Σουηδία ας πούμε. Ή όπου αλλού θέλει. Στην Ιταλία ξέρω εγώ. Υπάρχουν πάντως κέντρα αριστείας σε ορισμένες χώρες. Και αυτό μπορεί να το κάνει ο ασθενής εφόσον ενημερωθεί και διαγνωστεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τα, τα συμπτώματα λοιπόν πρέπει να είναι γνωστές τα, να είναι γνωστά συγγνώμη, τα συμπτώματα, τα πρώτα συμπτώματα στο τελευταίο χωριό της Ευρώπης, ώστε ο κόσμος να είναι ενημερωμένος. Στη δικιά μας την περίπτωση, εντάξει, η μητέρα μου δεν πέθανε από άνοια, ήταν στο νοσοκομείο, γιατί είχε μια πληγή και πέθανε τη νύχτα στο νοσοκομείο, γιατί υπήρξε κάποια δυσλειτουργία και δεν υπήρχε νοσοκόμος εκεί. Αλλά στο μεταξύ δεν θυμόταν ότι είχε πεθάνει ο πατέρας μου και η διαδικασία πήγε πάρα πολύ γρήγορα πρέπει να ξέρετε. Προχώρησε πάρα πολύ αρρώστια. Εγώ φρόντιζα βέβαια τη μητέρα μου, ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να μπορείς να βοηθήσεις τον άλλο να καταλάβει τι του συμβαίνει. Τις πρώτες βαμάδες που δεν θυμόταν Όταν έπαιρνα τηλέφωνο ή κάποιος της έλεγε «Κοίτα, στο τηλέφωνο είναι η κόρη σου, η Ντάγμαρ». Ε, ερχόταν στο τηλέφωνο, απαντούσε «Ναι», αλλά δεν είχε καταλάβει το «η κόρη σου» ή το όνομά μου. Μόνο όταν άκουγε τη φωνή μου καταλάβαινε ποια ήμουνα. Είναι και αυτό ένα σύμπτωμα. Πάντως, μέχρι την τελευταία μέρα καταλάβαινε ότι κάτι τη συμβαίνει και αυτό την τρόμαζε. Και γι' αυτό λέω ότι οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν τη διάγνωση, αλλά πρέπει συγχρόνω να ξέρουν και πώ μπορούν να βοηθηθούν. Δεν πρέπει να του πετάμε τη διάγνωση και τελείωσε. Όχι. Και γι' αυτό έχουμε αυτό το εργαστήριο. Ξέρω, εδώ συγκινούμε. Τι να κάνω, μιλάω για κάτι πολύ προσωπικό. Σα διηγήθηκα την ιστορία μου, γιατί η ιστορία μου δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μια καθημερινή ιστορία. Εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να σα πούν μια τέτοια ιστορία δεν συμβαίνουν μόνο μακριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβαίνουν πολύ κοντά μας όλο και περισσότερο. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε σήμερα να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κύριο Μπαρόσο και τους άλλους επιτρόπους να ξέρουν ότι θέλουμε τη στήριξή τους. Θέλουμε χρήματα για αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Αυτές είναι οι τελικές μου ε, τα τελευταία μου σχόλια. Τώρα έχουμε ένα σύντομο βίντεο. Έχουμε προσκαλέσει τον Ζαν εδώ πέρα. Οι περισσότεροι νομίζαν ότι θα έρθει όντω στην αίθουσα. Εγώ δεν ε, του είπα αμέσω αμέσω μπα, όχι. Σε βίντεο θα τον έχουμε. Αλλά και αυτό είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, το βίντεο. Boa tarde Μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλσχάιμερ και άλλες άνοιες ε, έχει υπερκομματικό χαρακτήρα, υπερβαίνει από την αρχή πάλι, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλσχάιμερ και άλλε άνοιε έχει υπερκομματικό χαρακτήρα. Υπερβαίνει τι ιδεολογικέ διαφορέ και τι διαφορέ ω προ τι σκεφτικέ πεπιθήσει. Δεν μπορούμε παρά να αποδώσουμε εύσημα σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Θα ήθελα να χαιρετήσω την Ομίγυρο, όλου του παρισταμένου βουλευτέ, εκπροσώπου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Συμβουλίου, όλου όσου ε, συμμετείχαν στο σημερινό εργαστήριο για να αναζητήσουμε από κοινού τι καλύτερε δυνατέ στρατηγικέ, ε, τι βέλτιστε λύσει, ε, ούτω ώστε να αντεπεξέλθουμε στη μεγάλη αυτή πρόκληση. Αναφέρομαι στου εκπροσώπους των ενώσεων των ασθενών, στου οικείου των ασθενών και στου ε, επαΐοντες που ήρθαν να καταθέσουν την μαρτυρία του ε, και να συμβάλλουν στη συζήτηση. Εγώ δέχτηκα την σημερινή πρόσκληση μέσω τη ε, βουλευτού Μαρίζα Ματίας για να συνταχθώ κι εγώ με τους υπόλοιπους αυτό τον αγώνα. Είναι τιμή μου και θέλω να δηλώσω αλληλέγγυο προ του ασθενεί, του πάσχοντε και του οικείου του. Ε, το να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης ε, των πασχόντων και των οικείων είναι μια μεγάλη πρόκληση και θα ήθελα να απευθύνω αυτή την ομιλία κυρίως σε αυτούς που βρίσκονται εγκύτερα στην ε, νόσο αυτή. Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σε αυτό το τομέα είναι ο σωστός δρόμος για να εγγυηθούμε ισότιμη πρόσβαση στις θεραπευτικές αγωγές για όλους, ισότιμη μεταχείριση ανεξάρτητα από τα εισοδήματά τους και από τον τόπο στον οποίο βρίσκονται. Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου και να εξημίσω την ελπίδα και το κουράγιο όλων όσων ε, υποφέρουν από την ε, νόσο του Αλχαέμι που πλήττει 8 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες ε, και κάθε χρόνο υπάρχουν 1,4 εκατομμύρια νέα κρούσματα και κάθε 20 χρόνια περίπου διπλασιάζει το αριθμός αυτός. Ένα νέο κρούσμα διαγιγνώσκεται κάθε 24 δευτερόλεπτα περίπου. Είναι τραγικό. Μιλούμε για αυτά τα νούμερα, για αυτά τα αριθμητικά στοιχεία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν μιλάμε για νούμερα μόνο. Μιλάμε για ανθρώπους, ε, για πραγματικές καταστάσεις. Ε, ε, πλήττεται η ζωή των ασθενών και των οικογενειών τους και γι' αυτό θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την νόσο, να βελτιώσουμε την ζωή των ασθενών και να αγωνιστούμε από κοινού. Γι' αυτό και εγώ θα ήθελα να συνταχθώ με όλους τους υπόλοιπους, ώστε να έχουμε τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Χρειάζεται ομαδική δράση ε, για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ε, μετά τη διάγνωση ε, δε της ενώσου θα πρέπει να κατοχυρώσουμε και την αξιοπρεπή διαβίωση των ασθενών. Πρέπει αυτό να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα. Μπορούμε να επιβραδύνουμε την εξέλιξη της νόσου αλλά όχι και να την ανασχέσουμε. Οπότε το μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα οφείλουμε να διατηρήσουμε την αυτονομία του ασθενού, να βελτιώσουμε τι συνθήκε διαβίωσή του και γνωρίζουμε ότι η εξάρτηση από τρίτου είναι κάτι αναπόφευκτο σε αυτή την νόσο ε, και ε, γι' αυτό θα πρέπει να ε, κατοχυρώσουμε επαρκείς συνθήκες ε, για όλους, να προσφέρουμε την κατάλληλη εκπαίδευση και ακόμη και αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας χρειάζονται και άλλες δράσεις από πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και εθνικές δράσεις για να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα. Εγώ είμαι αθλητής, είμαι επαγγελματίας στον τομέα του αθλητισμού και θέλω να υπενθυμίσω ότι η σωματική άσκηση είναι ένα σημαντικό παράγοντα ε, πρόληψη. Ε, λυπάμαι που δεν είμαι μαζί σα σήμερα, αλλά η ομάδα μου είχε αγώνα και χθε ε, και σε δύο μέρε. Ήταν αδύνατο να παραστώ στο εργαστήριο. Δηλώνω αλληλέγγυο πάντω και υποστηρίζω και του πάσχοντε και του οικείου του. Ευχαριστώ. However, you have done that, Marisa. Um, that will create a lot of support. That is. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις εντυπωσιακέ παρατηρήσεις του Ζαμορίνιο κλείνω το εργαστήριο. Θα δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η εισηγήτρια θα έχει να κάνει κάποιες προτάσεις επί της διαδικασίας. Μαρίζα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις εξαιρετικές παρεμβάσεις σας, όλες τις προτάσεις που κάνατε. Δεν έχουμε χρόνο, όντως, για να γίνει ανταλλαγή απόψεων, όπως είπατε κι εσείς. Παρόλα αυτά, θα ήθελα να κάνω κάποιες βασικές παρατηρήσεις. Γνωρίζετε όλο το περιεχόμενο της έκθεσής μου. Γνωρίζετε για ποιο πράγμα σας μιλώ. Θα ήθελα να παριθμίσω απλώς μόνο τα θεμελιώδη ζητήματα που πραγματευόμαστε μέσα στην έκθεση. Ε, και δεν, ε, αν λείπουν κάποια στοιχεία, ε, οφείλω να πω ότι περιορίστηκα ως προς την έκταση της έκθεσης, όχι επειδή δεν ήθελα να συμπεριλάβω όλα τα στοιχεία. συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά με όλους τους σκιώδεις εισηγητής και θα ήθελα τώρα να υπογραμμίσω το εξή. υποστηρίζω τους τέσσερις στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως το θέμα της πρόορης διάγνωσης και της πρόληψης, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια γιατί δεν γίνεται συντονισμένη προσπάθεια. Πρέπει να προωθήσουμε τα εθνικά ε, σχέδια δράσης ε, για να ε, υπάρξει και καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Γνωρίζετε επίση άλλου τομεί που αναφέρονται μέσα στην έκθεσή μου, έρευνα, παροχή περίθαλψης, θεραπευτικής αγωγής, ελάχιστη κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου, υποστήριξη προ τι οικογένειε των πασχόντων, παροχή καλή υπηρεσιών, ε, ισότιμη πρόσβαση για όλους τους ασθενείς ε, της νόσου Αλσχάιμερ. Αυτές είναι όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημά μας ε, και ε, χαίρομαι πάρα πολύ που ακούσαμε σήμερα τους εκπροσώπους των ασθενών. Ε, μπορώ να εμβαθύνω την ε, έκθεσή μου και φυσικά θα ξανασυναντηθούμε. Θα υπάρξουν και συνεδριάσεις για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε κύριε Ματία. Συγγνώμη που σας πιέζω, αλλά οι συνάδελφοι την έχουν διαβάσει την έκθεσή σας. Θα ήθελα για 1,5 λεπτό να δώσω την ευκαιρία και στους υπολείπους να μιλήσουν. και μετά ίσως να ξανακούσουμε τη Μαρίσα. Έχουμε δύο εναλλακτικέ λύσεις. Ε, είτε να αναβάλουμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια, αυτό δεν είναι θετικό για την Επιτροπή, ή ε, να ε, μείνουμε στο προανακοινωθέν χρονοδιάγραμμα, άρα δεν θα γίνει άλλη ανταλλαγή απόψεων. Θα συναντηθείτε εσείς με τους Κιώδης απλώς. Η Μαρίσα προτείνει να γίνει συνάντηση με τους Κιώδης πριν λήξει η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για συνεργαστούν. Κυρία Αντωνέσκου. Yeah, thank you very much. Uh, uh, θα ήθελα να χαρώ την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε για την έκθεση αυτή. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε το χρόνο πράγματι και ακριβώς γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω μόνο για την αναγκαιότητα μεγαλύτερης ε, ευαισθητοποίησης της κοινή γνώμης όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις. Μόλις ακούσαμε ότι το κάπνισμα έχει αρνητικές συνέπειες και μπορεί να επηρεάσει την ε, εξέλιξη της ασθένειας αρνητικά. Η κατανάλωση τροφίμων όπως τα ψάρια είπαμε ότι είναι κάτι θετικό. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο στις σχέσεις ανάμεσα στην έρευνα και την κοινή γνώμη αν θέλουμε να ελέγξουμε τελικά την αρρώστια. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω την ε, πολυδιάστατη μορφή του θέματος. Έχουμε την πρωτογενή έρευνα, έχουμε τη δημόσια υγεία, έχουμε την κοινωνική έρευνα, έχουμε τις υποστημενικές γνώσεις, οι οποίες πρέπει στην πράξη να ερμηνεύονται κλινικά. Αυτό είναι που έχει σημασία. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να δουλεύουμε στις διάφορες συναντήσεις που έχουμε οι συγητές μεταξύ μας. Και συμφωνώ να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Δανέσκου. Η κυρία Μακάβαν έχει τώρα το λόγο από τους σοσιαλδημοκρατές γιατί η κυρία Τσέση δεν είναι εδώ. Ναι, είναι άρρωστη, έπρεπε να φύγει. Είναι κρίμα που δεν είμαστε περισσότεροι εδώ. Το θέμα των ηλικιωμένων είναι ένα θέμα με το οποίο ερχόμαστε όλοι αντιμέτωποι κάποια στιγμή στη ζωή μας πρέπει να στηρίξουμε την Επιτροπή και τις προσπάθειές της. Μαρίσα, ευχαριστούμε για την έκθεση. Είναι πολύ καλή, πιστεύω. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη αρκετά πράγματα, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε και εδώ στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά. Να έχουμε ένα σχέδιο. Ίσως θα μπορούσαμε να επικεντρώσουμε την έκθεση περισσότερο σε αυτό. Μια αλλαγή που θα ήθελα να δω για παράδειγμα είναι κάτι για τη στήριξη της έρευνας ενδιατρικά. Πρέπει να στηριχτεί η έρευνα αυτή. Τα φάρμακα κοστίζουν ακριβά. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια τέτοια τροπολογία. Η κυρία Σίλτα θα ήθελε επίσης κάτι για τις λεγόμενες διαθήκες εν ζωή και την αναγνώρισή τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι άνθρωποι μετακινούνται. Μπορεί να έρθει ένας συγγενής από άλλη χώρα να πάει να ζήσει με έναν ασθενή. Θα πρέπει να μπορεί να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να αλλάξουμε την κατάσταση όσον αφορά την άνοια. Ας θέσουμε κάποιους στόχους λοιπόν. Φρεντερίκ Ρίς από τους Φιλελεύθερους. Η κυρία Ευχαριστώ. Ναι, μισή λεπτό έχω στην Ολομέλεια. Τέλος πάντων, σήμερα πιστεύω ότι η συζήτηση άξιζε τον κόπο, ακόμα και αν έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος για μας εδώ. Ζήσαμε συγκινητικές στιγμές, πράγματι. Θέλω και εγώ να ευχαριστώ όλους από το πάνελ που εμπλούτησαν τόσο πολύ τη συζήτησή μας. Τώρα σύντομα θα ξανασυζητήσουμε φυσικά με την εισηγήτρια την κυρία Ματιάς που ευχαριστώ. Ένα θέμα σχετικά με το οποίο εμείς ε, οι φιλελεύθεροι θέλουμε να γίνει κάτι παραπάνω είναι το εξή. Τι μπορεί να προσφέρει παραπάνω η Ευρώπη. Πέρα από αυτά που γίνονται στα κράτη-μέλη δηλαδή. Πέρα από τα σημεία 4 και 5 που μιλάνε για το συντονισμό και για τις προτεραιότητες των ε, κρατών μελών, πρέπει να υπογραμμίσουμε εμείς την έρευνα. Έρευνα για την ασθένεια του Αλσχάιμερ και γενικότερα για τις εκφυλιστικές ασθένειες. Έχω ερωτήσεις, διμερώς θα τις θέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συνέντευξη της κυρίας Ντατί στο περιοδικό Άνια, γιατί εκεί αναφέρει ένα σωρό προγράμματα τα οποία προβλέπονται στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για αυτό το τομέα. Θα ήθελα να ξέρω περισσότερα. Τι έχει γίνει στο προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο, για παράδειγμα. Αλλά θα το δω αυτό διμερώς. Τώρα, μια μικρή απόχρωση για το σημείο 9. Στο σημείο 9 η συγγήτρια μιλάει για την αμυλοειδή πλάκα και την αναφέρει σαν να είναι η μοναδική αιτία που προκαλεί το Αλσάιμερ όλοι συζητάμε με τους επιστήμονες και τους γιατρούς για αυτά. Οπότε, ίσως μαζί να πρέπει να το ξαναδούμε αυτό το σημείο. Έπειτα, η υπεραξία. Τι παραπάνω προσφέρει η έρευνα και η προτεραιότητα που δίνουμε στα δικαιώματα των ε, ασθενών. Παράγραφη 7, 8, 9, 11. Είναι ζωτική σημασία. Το ακούσαμε και η ε, καθηγήτρια Καπούτο και άλλοι είπαν ότι έχει πολύ σημασία να Ελαμβάνουμε υπόψη μας και τους περιθάλποντες. Και αυτό που είπαμε για τα κέντρα αριστείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω σε αυτό πρέπει να σκύψουμε παραπάνω. Ευχαριστούμε Φρεντερίκ, λέει Πρόεδρος. Η κυρία Χάσα έπρεπε να φύγει που είναι σκιώδης η από τους πρασίνους για ένα λεπτό. Μα πραγματικά ένα λεπτό, κύριε Ζουβά, ένα λεπτό. Ε? Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σε ένα λεπτό. Η έκθεση μπορεί να συμπληρωθεί πράγματι από μερικά σημεία. Πρώτον, μην ξεχνάμε τους νέους ασθενείς. Δεν είναι όλοι οι ηλικιωμένοι ασθενείς Αλσχάιμερ. Δεύτερον, για τα ιατρικοκοινωνικά μέτρα. Οι οικογένειες πώς μπορούν να βοηθηθούν να κρατήσουν τον ασθενή στο σπίτι. Τρίτον, έρευνα φυσικά και είναι θεμελιώδης, αλλά μην ξεχνάμε και την καινοτομία στην έρευνα. Μην επικεντρωνόμαστε σε ένα είδος έρευνας μόνο. Η καινοτομία πρέπει να είναι βασικό στοιχείο. Επίσης είναι σημαντικό να μιλήσουμε και για τη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γιατί εκεί λείπει πολλές φορές η καινοτομία. Τέλος, ηθική. Και αυτή πρέπει να συμπεριληφθεί σε μια τέτοιου έκθεση. Τίθενται και ηθικά ζητήματα με αυτή την ασθένεια. Ευχαριστούμε κύριε Ζουβέλη Πρόεδρος. Ναι. Τροπολογίες. Υποβάλλετε τροπολογίες. Προθεσμία είναι 9 Νοεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Όλοι οι σκιώδεις, παρακαλώ, και οι πολιτικές ομάδες που δεν έχουν εδώ σκιώδεις και πράσινα δηλαδή, και της κυρίας Γιανακουδάκη ομάδα, να ξέρετε ότι προβλέπει η κυρία Μάτιας πριν την λήξη της προθεσμίας μια συνάντηση με τους Κιώδης. Δευτέρα, 8 του μηνός. Εμείς ξεκινάμε την Τρίτη το πρωί στις 9 με ψηφοφορίες. Άρα 8 η ώρα το βράδυ θα είσαστε όλοι στις Βρυξέλλες. Μπορείτε να πάτε σε αυτήν, στη... στις 8 του μηνό, συγγνώμη, θα είσαστε όλοι. Κατά τις 5 μάλλον θα λάβει χώρα η συνάντηση αυτή με τους Σκιώδης. Φροντίστε να είσαστε 8 του μηνό. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών. Είπαμε 9 του μηνό, 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Έληξε το εργαστήριο αυτό. Η εισηγήτρια για τον τελευταίο λόγο. Ευχαριστώ. Δύο λόγια έχω να πω. Αλλά δεν θα τα πω τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ και όλους τους συμμετέχοντες για την τόσο ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Υπογραμμίζω για άλλη μια φορά αυτό που ακούσα από την κυρία